Secretary. Το θυμάστε.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 Allora, colleghi, il servizio dovrebbe di... Λοιπόν, από ό,τι φαίνεται λέει η Πρόεδρος, το σύστημα λειτουργεί πάρα πολύ ωραία λοιπόν. Μπορούμε να ξαναρχίσουμε τις εργασίες μας. Το επόμενο σημείο της σημερισίας διατάξεως είναι η ψηφοφορία επί δύο θεμάτων. Το ένα είναι το σημείο 10, γνωμοδέτη για τις κατευθυντήρες γραμμές του προϋπολογισμού για το 2012 πριν από την ψηφοφορία έχουμε την κυρία Ούκηνη, η οποία έχει δει το λόγο. Ναι, πολύ σύντομα. Σχετικά με το διαμεσολαβητή θέλω να κάνω μια αναφορά. Είναι εξαίρετη αυτή η έκθεση. Όμως νομίζω θα πρέπει να σκεφτούμε ότι εάν ο διαμεσολαβητής ε, ε, έμενε στο Στρασβούργο θα γλιτώναμε πάρα πολλά χρήματα γιατί πάρα πολύ κόστος αφορά τα ταξίδια, τις μετακινήσεις κτλ. Νομίζω λοιπόν ότι πρέπει με κάποιο τρόπο να βελτιώσουμε την κατάσταση αυτή όσον αφορά τον διαμεσολαβητή. Ε, να έρθουν στις Βρυξέλλες μάλλον, στις Βρυξέλλες. Και έτσι θα κερδίζαμε πάρα πολλά ε, χρήματα. Ευχαριστώ. Θέλει κάποιος άλλος το λόγο. Όχι από ό,τι φαίνεται. Επομένως ξεκινάει η συζήτηση, η ψηφοφορία, συγγνώμη. <clears throat> Τροπολογία 1, παράγραφος 1, υπέρ κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 2 στον παράγραφο 2, υπέρ, κατά, εγκρίνεται. Τροπολογία 3, παράγραφος 3, υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Τροπολογία 4. Για την τροπολογία 4 προβλέπεται και προφορική τροπολογία εν είδη τεχνικής διορθώσεως. Συμφωνούν όλοι, ωραία, επομένως ψηφίζουμε την τροπολογία 4 παράγραφος 5 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 5 επί της παραγράφου 5 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 6 επί της παραγράφου 7 υπέρ κατά αποχές. Δεν είναι σαφές το αποτέλεσμα. Μπορούμε να επαναλάβουμε την ψηφοφορία, παρακαλώ. Υπέρ. Τροπολογία 6 επί της παραγράφου 7. Υπέρ. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Αποχές, συγγνώμη λέει η πρόεδρος, το ξέχασα, εγκρίνεται. Τροπολογία 7 επί της παραγράφου 8α υπέρ. Κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τελική ψήφος υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Ετήσια έκθεση για τον Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή πριν αρχίσει η ψηφοφορία. Θέλει κάποιος να πάρει το λόγο. Παρακαλώ. Uh, because I am replacing την κυρία Ιώτοβα σήμερα. Θα ήθελα να ευχαριστήσει όλους όσους συνεργάστηκαν στην ε, σύνταξη της, της γνωμοδότησης. Είχε μια εξαιρετική ε, συνεργασία και αυτό είχα να πω μόνο εκ μέρους της. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ, λέει η Πρόεδρος. Επομένως ξεκινάει η ψηφοφορία. Τροπολογία 9 της παραγράφου 2α υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 10 της παραγράφου 7α υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 11 επί της 8α υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 12 παράγραφος 9 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 13 επί της παραγράφου 9α υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 14 επί της παραγράφου 11α υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 15 επί της παραγράφου 12 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 16 επί της παραγράφου 13 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Συμ... Συμβαστική τροπολογία Β υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Οι 17 και 18 καταπίπτουν. Τροπολογία 19 της παραγράφου 15 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 20 από της παραγράφου 16 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 21 από της παραγράφου 18 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 22 επί της 18α υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 23 επί της παραγράφου 19 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 24 επί της παραγράφου 20 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική τροπολογία C, γάμα, επί της παραγράφου 21 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Καταπίπτουν οι τροπολογίες 25, 20, 26, 27 και 28. Περνάμε στην τροπολογία 29 για το 22α. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 30, παράγραφος 22α. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Περνάμε τώρα στα αιτιολογικά. Τροπολογία 2 επί του α υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 3 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 4 με μία διόρθωση τεχνικής φύσεως. Ε, δεν αντιτίθεται κανείς αυτή τη διόρθωση, όχι, επομένως ψηφίζουμε το 4, έτσι όπως έχει τροποποιηθεί, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 5, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβιβαστική τροπολογία α, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 6 και 7 καταπίπτουν, φτάνουμε στην τροπολογία 8, υπέρ, κατά, επαλήθευσης. Ψηφίζουμε λοιπόν την τροπολογία 8 εκ νέου επί του H α υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 1 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τελική ψηφοφορία υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Σας ευχαριστώ πολύ. Ολοκληρώθηκαν οι ψηφοφορίες και περνάμε λοιπόν στο επόμενο σημείο της ημερησίας διατάξεως. Πρόκειται για μια ε, προκαταρτική αναφορά όσον αφορά τη διερευνητική επίσκεψη στη Βουλγαρία. Επί του σημείου, κύριε Σαλαβράκο. Ε, όχι, θα, θα παρακαλούσα να διευκρινιστεί. Θα παρακαλούσα να διευκρινιστεί εάν θα πάμε στη Ρουμανία και ποιες ημερομηνίε για να έχουμε το χρόνο να, να απαντήσουμε διότι μέχρι το Σεπτέμβριο που θα το ξανασυζητήσουμε το θέμα είναι αρκετός ο χρόνος. Να δούμε πότε ακριβώς μπορούμε να πούμε ναι ή όχι. Για τη Ρουμανία, για το Βουκουρέστι. Αγαπητέ συνάδελφε, αποφασίστηκε και εγκρίθηκε η επίσκεψη στη Ρουμανία. Οι ημερομηνίε ακόμα δεν έχουν επιβεβαιωθεί. Θα πάμε σίγουρα, δεν ξέρουμε όμω ακόμα πότε. Επομένω, περνάμε στο επόμενο σημείο, σημείο 12, ε, έκθεση όσον αφορά τη διερευνητική επίσκεψη στην Βουλγαρία. Θα έχουμε μια πρώτη πληροφόρηση. Η κυρία Όουκεν θα μας την κάνει, θα μας την δώσει. Dansk. Θα ήθελα να μιλήσω δανέζικα, είναι δυνατόν. Βεβαίως. Put on your earphones. Θα μιλήσω δανέζικα λοιπόν. Eh, eh, Ωραία. Λοιπόν, Όπως είπαμε χτες, αποφασίσαμε να επισκεφθούμε διάφορα, ε, να κάνουμε διάφορες επισκέψεις βάσει αυτών που μας πρότεινε ο κ. Κωστινά. Jeg var alene. Victor havde sagt fra begyndelsen, Είπαμε λοιπόν ότι ε, η επίσκεψή μας ήταν ε, ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα. Θα μπορούσα να σας δώσω βέβαια πολλές πληροφορίες αυτή τη στιγμή. Είδαμε πάρα πολλά πράγματα. Είδαμε ποια είναι τα προβλήματα τα οποία αυτή τη στιγμή αντιμετωπίζει η χώρα αυτή. Στην πρώτη συνάντηση που είχαμε με τον δήμαρχο της πόλης της Σόφιας, συζητήσαμε για το ζήτημα του Σολοντόρ. Έγινε μια ανταλλαγή απόψεων μαζί με διάφορους αναφέροντες, μαζί με τις τοπικές αρχές. Προσπαθήσαμε λοιπόν να συμβάλλουμε στην ε, επίλυση των προβλημάτων που έχουν παρουσιαστεί. Είχαμε έντονες συνομιλίες, όπως σας είπα, με τον ε, Δήμαρχο και είδαμε ότι όντως υπήρχε ένα πολύ σημαντικό πρόβλημα με τη συγκεκριμένη χωματερή. Γνωρίζω ότι υπάρχει μια γνωμοδότηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής όσον αφορά τη διάθεση των απορριμμάτων στο, στην περιοχή αυτή. Δεν γνωρίζαμε όμως εμείς την γνωμοδότηση αυτή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής όταν πήγαμε στη Βουλγαρία. Το... Είδαμε το κείμενο αυτό μόνο μετά την επιστροφή μας Πήγαμε πάντως στη χωματερή αυτή, είναι τεραστίων διαστάσεων, καλύπτει ένα πολύ μεγάλο γεωγραφικό, γεωγραφική απόσταση. Βρίσκεται πολύ κοντά στην πόλη της Σόφιας και προφανώς προκαλεί προβλήματα στην πόλη της Σόφιας. Πήγαμε λοιπόν το Σάββατο στην χωματερία αυτή, επί τόπου ήταν και οι αναφέροντες, αλλά και ο διευθυντής της εταιρείας που διαχειρίζεται τη χωματερή αυτή, Υπήρχαν επίσης πάρα πολλά φορτηγά. Υπήρχε μια έντονη δραστηριότητα, πάντως μας είπαν τόπου ότι όλα αυτά ήταν ένα τεράστιο ψέμα. Ότι ειδικά για μας, για την επίσκεψή μας στη χωματερία αυτή, είχαν κινητοποιήσει όλους αυτούς τους φορείς. Μας εξήγησαν ότι στην πράξη τα πράγματα δεν λειτουργούν έτσι. Σκηνοθετήθηκε λοιπόν, αν θέλετε, όλη αυτή η υποτιθέμενη δραστηριότητα σε αυτή τη χωματερή μόνο και μόνο για να εντυπωσιαστούμε εμείς στα πλαίσια της αποστολής μας. Πιστεύω λοιπόν ότι στην περίπτωση αυτή του Σοροντόλ στην Βουλγαρία θα πρέπει να γίνει κάτι. Θα πρέπει να ασχοληθούμε ακόμα περισσότερο προκειμένου να επιλύσουμε όλα τα προβλήματα που έχουν να κάνουν με την διάθεση των απορριμμάτων. Συζητήσαμε επίσης με τον ε, αρμόδιο υπουργό στη Βουλγαρία, ο οποίος ε, μας παρουσίασε τα πράγματα εντελώς ιδηλιακά. Μας είπε ότι ε, όλα λειτουργούν άψογα. Είχαμε σχεδόν την εντύπωση ότι βρισκόμασταν σε μια κομμουνιστική Βουλγαρία, όπου οι επίσημες αρχές μας λέγανε ότι τα πάντα λειτουργούν πάρα πολύ θετικά και ότι δεν παρουσιάζεται κανένα απολύτως πρόβλημα. Έτσι παρουσίαζαν λοιπόν τα πράγματα οι εκπρόσωποι τη κυβέρνηση όσον αφορά την ε, διαχείριση και την προστασία του περιβάλλοντο. Εντελώ διαφορετική εικόνα βέβαια είχαμε όταν μιλήσαμε με τον επικεφαλή Επιτροπή Αναφορών του ε, Βουλγαρικού Κοινοβουλίου και όταν μιλήσαμε και με τον διαμεσολαβητή του, της Βουλγαρίας, τον συνήγορο του πολίτη, η οποία μας παρουσίασε τα πράγματα βέβαια εντελώς διαφορετικά από μια άλλη σκοπιά, από μια άλλη οπτική γωνία. Πρέπει να σας πω επίσης ότι στο παρελθόν ο συνήγορος του πολίτη διοριζόταν άμεσα από το κυβερνόν κόμμα, πράγμα το οποίο δεν συμβαίνει αυτή τη στιγμή και πράγμα το οποίο είναι αδιανόητο για ορισμένε χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης, ιδίως για τις ε, βόρειες χώρες. Είχαμε επίση στο Ριλεμπιέν, όπου είναι ένα από τα πιο σημαντικά ενδιατήματα στην Ευρωπαϊκή Ένωση ένας από τους πιο σημαντικούς οικότοπους. Και πηγαίνοντας προς την περιοχή αυτή, μας είπαν ότι στον, στην περιοχή αυτή προσπαθούν να δημιουργήσουν αυτή τη στιγμή ένα τεράστιο ολικό πάρκο και ότι αυτό ουσιαστικά θα επηρεάσει πάρα πολύ τη ζωή των πτηνών κυρίως που ζουν στον βιότοπο αυτό, στον οικότοπο αυτό. και από ό,τι φάνηκε δεν γινόταν ε, σεβαστή νομοθεσία του Natura 2000 για τη συγκεκριμένη αυτή περιοχή στη Βουλγαρία, στα πλαίσια δηλαδή των κατασκευαστικών σχεδίων για το τεράστιο αυτό ελικό πάρκο το οποίο ε, θα δημιουργηθεί. Είναι πάρα πολύ σημαντικό λοιπόν στα πλαίσια της αδειοδότησης της δημιουργίας αυτού του υλικού, αφού πάρκου να ληφθούν υπόψη όλες οι προδιαγραφές και όλοι οι κανόνες που ισχύουν στα πλαίσια του Natura 2000. Πήγαμε επίσης σε ένα χιονοδρομικό κέντρο. Και προς αυτό είχαν υποβληθεί κάποιες αναφορές. Οι αναφέροντες θέλαν να εξασφαλίσουν ότι από τεχνικής πλευράς τα πράγματα θα, θα εξελιχθούν ομαλά, ότι το χιονοδρομικό αυτό κέντρο και η κατασκευή του δεν θα επηρεάσουν το περιβάλλον οι αναφέροντες ε, παρουσίασαν μια σημαντικότατη τεκμηρίωση. Επίσης μας είπαν ότι ε, ήταν πολύ δύσκολη η πρόσβαση στην περιοχή αυτή γιατί θεωρείται ως ε, ιδιωτική ιδιοκτησία ενώ κανονικά η έκταση αυτή θεωρείται δημόσιο αγαθό, δημόσια ιδιοκτησία. Υπάρχουν ε, πάρα πολλοί άνθρωποι που επισκέπτονται την περιοχή αυτή, την περιοχή του χιονοδρομικού κέντρου, που κανονικά και αυτή υπάγεται στα πλαίσια του Natura 2000. Έχει γίνει ένας τεράστιος πόλος έλξης για πάρα πολλούς ε, τουρίστες και δεν θα πρέπει να ξεχνάμε βέβαια ότι είναι κανονικά μια προστατευόμενη περιοχή στην οποία ζουν πάρα πολλά πτηνά. Όταν ε, φτάσαμε στο χιονοδρομικό αυτοκέντρο κέντρο είδαμε ότι υπήρχαν και εκπρόσωποι από τον εκεί Δήμο, από τις τοπικές αρχές Είχε διοργανωθεί μια πολύ μεγάλη διαδήλωση από τους πολίτες. Αποφασίσαμε τελικά να μην πάμε στο συγκεκριμένο αυτό τόπο, γιατί δεν θέλαμε σε καμία περίπτωση να δώσουμε την εντύπωση ότι συμμετέχουμε κι εμείς άμεσα στην ε, διαδήλωση αυτή. Για μια δεύτερη πάντως φορά καταφέραμε να δούμε πώς ε, οι τοπικές αρχές μαζί με διάφορους επιχειρηματίες προσπαθούν να δώσουν μια ψευδή εικόνα των πραγμάτων. να πω κάτι ακόμα στον αφορά το τμήμα αυτό της επίσκεψής μας. Ο δήμαρχος της εκεί περιοχής ε, μας είπε ότι ε, η κοινοτική νομοθεσία δεν ήταν μια απόλυτη προτεραιότητα για αυτόν. Το σημαντικότερο για αυτόν ήταν η ολοκλήρωση των κατασκευαστικών έργων και η προώθηση του τουρισμού. Αυτή ήταν η μόνη του μέρημνα και μάλιστα ακολουθούσα, θέλετε, κάποιες πεπαλαιωμένες πλέον προσεγγίσεις όσον αφορά τον ε, τουρισμό. Θεωρούσε ότι η δημιουργία μεγάλων εγκαταστάσεων θα προσελκούσε περισσότερους τουρίστες, χωρίς να συνειδητοποιεί ότι η προστασία του περιβάλλοντος μπορεί να λειτουργήσει εξίσου θετικά. Για να δημιουργηθεί λοιπόν το εθνοδρομικό αυτό κέντρο, καταστράφηκε ένα μεγάλο τμήμα της προστατευόμενης περιοχής, χρειάστηκε να κοπούνε πάρα πολλά δέντρα, οι αρχές βέβαια προσπάθησαν να το δικαιολογήσουν αυτό, λέγοντας ότι ε, στις περιοχές όπου κόπηκαν τα δέντρα αυτά θα προωθούνταν διάφορες καλλιέργειες για σημαντικά αγροτικά προϊόντα. Και ανάλογα παραδείγματα είχαμε και αργότερα κατά τη διάρκεια της ε, αποστολής μας σε άλλες περιοχές της ε, χώρας. Σε κάθε περίπτωση αυτό που είδαμε είναι ότι οι τοπικές αρχές προσπαθούν να χρησιμοποιήσουν κάποιες προστατευόμενες περιοχές προκειμένου να δημιουργήσουν χώρους για φεστιβάλ. Μας είπε για παράδειγμα ο Δήμαρχος ότι ένα πολύ σημαντικό φεστιβάλ jazz ή rock αν θέλετε θα λάμβανε χώρα σε αυτή την περιοχή. Είδαμε λοιπόν ότι πάνω στο βουνό αυτό θα διοργανώνταν αυτό το φεστιβάλ και προκειμένου να διοργανωθεί το φεστιβάλ αυτό είχαν δημιουργηθεί απαραίτητες εγκαταστάσεις οι οποίες βέβαια αντιτίθενταν σε κάθε μέτρο προστασίας του περιβάλλοντος και από την περιοχή αυτή βέβαια είχε, κάποιο, είχε κανείς μια καταπληκτική θέα προς τη γύρω φύση. Όταν θίξαμε το ζήτημα αυτό των μεγάλων αυτών εγκαταστάσεων στη φυσική αυτή περιοχή, προσπάθησαν οι τοπικές αρχές να δικαιολογήσουν κάπως την στάση τους, αλλά δεν κατάφεραν να μας πείσουν. Ανάλογα παραδείγματα είδαμε και σε άλλες ορεινές περιοχές της Βουλγαρίας, όπως το Περνίγκ για παράδειγμα, που και εκεί πάλι υπάρχει ένα χιονοδρομικό κέντρο, και όπου και εκεί πάλι είχε γίνει μία προσπάθεια από τις τοπικές αρχές να μας παρουσιάσουν μία ψευδή οροποιημένη εικόνα των πραγμάτων. Μας πρότεινε επίσης να διοργανώσουμε μία συνέντευξη τύπου πριν, κατά διάρκεια ή μετά την επίσκεψή μας. Ε, στόχος μας δεν ήταν σε καμία περίπτωση να διοργανώσουμε εμείς μία συνέντευξη τύπου, ιδίως κατά τη διάρκεια μίας ε, διαδήλωσης. Εμείς σε κάθε περίπτωση προσπαθήσαμε να μην εμπλακούμε σε καμία περίπτωση εσωτερικής διαμάχης στην Βουλγαρία. Και πάλι είδαμε ότι κάθε φορά που ήταν παρούσες οι τοπικές αρχές, δίπλα τους βρίσκαμε και διάφορους εκπροσώπους επιχειρήσεων ή φορέων εκμετάλλευσης. και είδαμε ότι οι περισσότεροι φορεί εκμετάλλευση ουσιαστικά έχουν προχωρήσει ένα καθεστώ joint venture μαζί με τι τοπικέ αρχέ. Και αν θέλετε να πούμε τα πράγματα και λίγο διαφορετικά, μπορούμε να πούμε ότι υπάρχει ένας πολύ μεγάλος βαθμός, ένα πολύ ψηλό επίπεδο διαφθοράς. Στη σύμπραξη αυτή που εμφανίζεται τελικά να είναι πάρα πολύ συχνή ανάμεσα στους τοπικούς επιχειρηματίες και φορείς εκμετάλλευσης και τις τοπικές αρχές. Πολλές φορές έχουμε δει ότι η δημόσια υπηρεσία ιδιωτικοποιείται και αυτό γίνεται προς όφελος τόσο των επιχειρηματιών όσο και των εκπροσώπων τοπικών αρχών πραγματικά ουσιαστικά υπάρχουν σημαντικότητα οικονομικά συμφέροντα τα οποία καθοδηγούν τις επιλογές που γίνονται από τις τοπικές αρχές και τους επιχειρηματίες. Όσον αφορά λοιπόν τέτοιες συμφωνίες joint ventures έχουν υποβληθεί από βούλγαρους πολίτες διάφορες αναφορές. Εμείς ως Επιτροπή αναφορών δεν μπορούμε να κάνουμε έρευνες, μπορούμε απλώς να ακούσουμε τα διάφορα σχόλια, μπορούμε να θέσουμε κάποιες ερωτήσεις, αλλά δεν μπορούμε να κάνουμε επίσημα κάποια έρευνα όσον αφορά τα γεγονότα αυτά. Καταλαβαίνετε ότι ασχολούμαστε πολύ συχνά με την Natura 2000, αλλά θεωρώ ότι τα ζητήματα αυτά ουσιαστικά ξεπερνούν τις αρμοδιότητές μας. Υπάρχει ένα ουσιώδες λάθος που είναι ε, ε, σφάλμα και πρόβλημα, που είναι η έλλειψη διαφάνειας. Το έχω συζητήσει και με άλλους συναδέλφους αυτό. Ε, οι αρχές ε, βεβαίως περηφανεύονται ότι υπάρχει πολύ μεγάλη διαφάνεια, αλλά εμείς επί τόπου διαπιστώσαμε ότι πόρο απέχει η διαπίστωσή μας από την ε, εξαγγελία των αρχών. Η δυνατότητα παρέμβασης των πολιτών είναι πολύ ή μάλλον θα έλεγα υπερβολικά περιορισμένη. Πρέπει να υπάρχει ε, ε, και πρέπει να, να καταλάβουμε ότι εάν δεν ε, αναλυφθεί δράση και από πλευρά των πολιτών και αν οι πολίτες δεν αναμειχθούν ενεργά στη διαδικασία, δεν θα υπάρξει ποτέ ένα καλό αποτέλεσμα. Η Βουλγαρία πρέπει να είναι περήφανη για αυτό το δίκτυο κοινωνικής συμμετοχής, αυτό το δίκτυο συμμετοχής των πολιτών βλέπουμε και γνωρίζουμε και υπάρχει και η σχετική τεκμηρίωση ότι οι πολίτες της Βουλγαρίας ενδιαφέρονται ενεργά και επομένως θα πρέπει να αναμειχθούν και με μεγαλύτερη διαφάνεια, κάτι το οποίο δεν διαπιστώσαμε στην Βουλγαρία. Νομίζω ότι μπορώ να ολοκληρώσω, δεν νομίζω ότι έχω κάτι άλλο. Και η Μαρία ήταν μαζί μας και την ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συμμετοχή της. Είχαμε την ε, δυνατότητα επίσης ε, να ε, ζήσουμε έτσι λίγο το τοπικό πνεύμα και αν ξέχασα κάτι, άλλοι συνάδελφοι θα ήθελα να με βοηθήσουν να καλύψουμε το πρόβλημα. Ευχαριστούμε πολύ και η συνάδελφε Όκεν, λέει η Πρόεδρος. Είναι γεγονός ότι η αποστολή αυτή σιγά σιγά φιλορώησε όσον αφορά την συμμετοχή. δίνω το λόγο στον κύριο Μποστινάρου. Ευχαριστώ πολύ αγαπητή Πρόεδρε. Θα ήθελα να <laughs> μιλήσω στη μητρική μου γλώσσα, στα ρουμανικά, όπως έκανε και η Μάργαρετ προηγουμένως. Σα πρέπει να πούμε ότι δεν είναι δυνατόν να αλλάζει η σύνθεση της αντιπροσωπείας που επισκέπτεται μία χώρα ε, τελευταία στιγμή και χωρίς να υπάρχει δυνατότητα ε, πρώτερης συζήτησης και με τις πολιτικές ομάδες, γιατί μπορεί να δημιουργηθεί δυσπιστία στην Επιτροπή μας. Δεύτερον, και αυτό είναι ένα μήνυμα πάλι για τη γραμματεία, δεν πρέπει να αλλάζει τελευταία στιγμή η ημερήσια διάταξη. Η ημερήσια διάταξη αποτελεί αντικείμενο συμφωνίας. Δεν μπορεί τελευταία στιγμή να αλλάζει. Όσον αφορά τώρα την ίδια την αντιπροσωπεία. Δηλαδή την ίδια την αποστολή θέλω να πω. Συμφωνώ με την κυρία Όκεν και είμαι πεπισμένος ότι η γραπτή έκθεση που θα βασίζεται στο σύνολο των συνεισφορών θα παρουσιάσει τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της επίσκεψής μας στη Βουλγαρία. Θα ήθελα ε, όμως να υπογραμμίσω κάποια στοιχεία τα οποία μου φαίνονται σημαντικά. Διαφάνεια έλλειψη διαφάνειας, αλλά και έλλειψη θεσμοθετημένου διαλόγου μεταξύ των ενδιαφερομένων μερών είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Έλλειψη διαλόγου μεταξύ μη κυβερνητικών οργανώσεων και υπουργείων. Έλλειψη διαλόγου ανάμεσα στους πολίτες και τις τοπικές αρχές. Ε, διάλογος με ανθρώπους ε, οι οποίοι οφείλουν να εκφράσουν τη γνώμη τους ε, επί ενός δεδομένου σχεδίου. Παντελής λοιπόν έλλειψη διαλόγου. Σε περίπτωση ε, παραβίασης ε, είτε της νομοθεσίας της Βουλγαρίας είτε της ε, ευρωπαϊκής νομοθεσίας θα πρέπει οπωσδήποτε να υπάρξει διάλογος ώστε να αποφευχθεί παρανόησης ή και διαμάχη. Στην Σόφια πρώτη φορά η πρώτη συνάντηση που έγινε μεταξύ των αρχών και των ε, ε, αναφερόντων ήταν με την ευκαιρία της επίσκεψής μας στη Βουλγαρία. Επομένως πρώτο μας μέλημα και πρώτο μας βήμα και αυτό είναι και ένα μήνυμα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, ενίσχυση του διαλόγου. Θα πρέπει και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να ασκήσει οποιαδήποτε πίεση έτσι ώστε να διασφαλιστεί ο θεσμικός διάλογος ανάμεσα στις αρχές ε, και την κοινωνία των πολιτών πρέπει αυτή η διασύνδεση να λάβει χώρα και εσείς σαν Ευρωπαϊκή Επιτροπή να βεβαιωθείτε ότι υπάρχει ο διάλογος αυτός σε τοπικό επίπεδο. Δεν πρέπει να, ε, να εξαπατώνται οι πολίτες. Δεύτερο στοιχείο όταν συναντήσαμε την Υπουργό Περιβάλλοντος, η κυρία Υπουργός μας έκανε μία σωστή παρουσίαση, η οποία ανεφέρεται στο νομικό πλαίσιο και αποκομίσαμε γενικά θετικές εντυπώσεις. Όμως, δύο πράγματα μας εξέπληξαν αρνητικά. Πριν από την επίσημη συνάντηση, η βουλγαρική κυβέρνηση μιλούσε για την νομιμοποίηση αναπτυξιακών προγραμμάτων στα ε, όρη της Ρίλα και του Ρούντοκ. Δηλαδή νομιμοποίηση ε, κάποιων παρανομιών και παρανόμων διαδικασιών. Και στην ουσία Αυτά που ακούσαμε μετά από την ε, ε, Υπουργό και αυτά που ξέραμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ήταν απολύτως ε, αντίθετα από αυτά που ακούγαμε επί τόπου όσον αφορά αυτή την νομιμοποίηση. Επομένως, τρανό παράδειγμα ε, που άλλα λέγονται και άλλα πράττονται μιλάμε εδώ για υποδομές οι οποίες οικοδομήθηκαν με ε, είτε παράνομους τρόπους, είτε στα όρια της νομιμότητας, άρα και στα όρια της παρανομίας, και μιλάμε για περιοχές οι οποίες εμπίπτουν στην ε, Natura 2000 ε, και για τις οποίες υποτίθεται ότι έπρεπε να έχουν γίνει μελέτες, περιβαλλοντικών επιπτώσεων και εν πάση περιπτώσει μιλάμε για περιοχές για τις οποίες ε, το φυσικό κάλος είναι σημαντικό και επομένως και οι επιπτώσεις από περιβαλλοντική άποψη είναι πάρα πολύ σημαντικές. Ε, πρέπει να δούμε λοιπόν, ε, ζητήσαμε ε, να μάθουμε ποιοι ήταν οι υπεύθυνοι για την αδειοδότηση αυτών των έργων. Συναντήσαμε λοιπόν τον δήμαρχο της περιοχής και μας είπε λοιπόν ότι για την περίπτωση των ε, ε, οροσυρών ε, ρίλα εκεί υπήρχαν οι απαραίτητες αδειοδοτήσεις αλλά στην ουσία είδαμε ότι στα όρη ρίλα τα πράγματα δεν ήταν έτσι όπως έπρεπε να είναι. Μιλάμε για υποδομές οι οποίες ξεκίνησαν να οικοδομούνται το 1995 και οι οποίες μπορεί να είχαν στην αρχή μια νόμιμη βάση αλλά σιγά σιγά έβριθαν παρανομιών. Και εκεί ε, εφαρμόστηκε η αρχή, αφού έγινε τώρα δεν μπορεί να ξεγίνει. οι τοπικές και περιφερειακές αρχές επανελάμβαναν διαρκώς ότι υπήρξαν σημαντικές μελέτες όσον αφορά την προστασία του περιβάλλοντος στα πλαίσια της Natura 2000. Μας είπαν ότι η πρόσβαση ήταν περιορισμένη, ότι ο αριθμός των επισκεπτών ήταν περιορισμένο, αλλά εμείς βλέπαμε ε, την ε, αναντιστοιχία των λεγόμενων με αυτά που έβλεπαν τα μάτια μας. Βλέπαμε να περνούν αυτοκίνητα ε, με τουρίστες, βλέπαμε μάλιστα και πούλμαν τουριστών που μετέφεραν... και και επίσης ε, μετέφεραν και εκατοντάδες, ε, ε, εκατοντάδες πολιτών που υποτίθεται ότι στήριζαν ενθουσιοδός το έργο. Θα δείτε και φωτογραφίες για να καταλάβετε, θα, δείτε, θα υπάρχουν και φωτογραφίες στην έκθεση για να καταλάβετε πώς είναι τα πράγματα. Είναι δεκάδες οι άνθρωποι οι οποίοι λούονται την θερινή περίοδο σε αυτές τις ε, λίμνες. Τέλος. Τέλος λέω. 145.000 ε, πολίτες ε, έχουν υπογράψει την ε, συγκεκριμένη αναφορά και έχουν υποβληθεί και άλλες δύο αναφορές. Και βεβαίως εγώ εντυπωσιάστηκα από την ισχυρή δέσμευση αυτών των ανθρώπων αλλά και την τεκμηριωμένη παρουσίαση των αναφορών. Το, η επιστημονική παρουσίαση καταδεικνύει ότι μονάχα 12 άνθρωποι θα πρέπει ταυτοχρόνως να εισέρχονται σε αυτήν την περιοχή έτσι ώστε να την προστατεύσουμε πραγματικά. Και εγώ είδα εκατοντάδες επισκέπτες. Και στρεφόμενος και προς την Επιτροπή πρέπει να πω ότι ε, η προσέγγιση της Επιτροπής ήταν λίγο αθώα και λίγο ιδεαλιστική. Γιατί πραγματικά τα γεγονότα μιλούν από μόνα τους. Τα στοιχεία καταδεικνύουν ότι τα πράγματα δεν είναι έτσι όπως τα έχουν παρουσιάσει. Και επομένως πρέπει να δράσουμε. Και τέλος, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε περιπτώσεις που έχουν τέτοιο βαθμό ευαισθησίας, ε, σε περιπτώσεις όπου τόσο, τόσοι πολλοί Ευρωπαίοι πολίτες αναφέρουν ένα πρόβλημα θα πρέπει να βρει τους μηχανισμούς και τα εργαλεία που θα ε, ε, επιτρέψουν να επαληθεύονται ή ε, να υπελθεύεται η ορθότητα των πληροφοριών και των στοιχείων που από τις κυβερνήσεις, από τις χώρες αυτές, είτε αυτές, αυτή είναι η Γερμανία, είτε είναι η Ρουμανία, είτε οποιαδήποτε άλλη χώρα, ότι λέω οι πληροφορίες αυτές είναι ορθές, θα πρέπει να ελέγχεται η ορθότητα. Εν πάση περιπτώσει, Στη διάρκεια της επίσκεψής μας ε, στην ε, Ρίλα, ε, εμείς διαπιστώσαμε ότι έγινε προσπάθεια να ασκηθεί πίεση, ας πούμε τα πράγματα με το όνομά τους, να ασκηθεί πίεση σε μια αντιπροσωπεία του Κοινοβουλίου. Αυτό είναι, το ελάχιστο μπορώ να πω, περίεργο. Ο υπεύθυνος της διαδικασίας στην ουσία ε, ενθάρρυνε, παρότρινε τους παρισταμένους να διαμαρτυρηθούν κατά της αντιπροσωπείας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Και αυτό το βρήκα πραγματικά παράτερο. Θα πρέπει κάποιος να εξηγήσει στους ανθρώπους αυτούς ότι η Ευρώπη προσπαθεί να τους προστατέψει. Και ότι ε, έχει η Ευρώπη κάποιους κανόνες, οι οποίοι κανόνες όμως αγνοούνται πλήρως. Τελευταία παρατήρηση. Ε, χαίρομαι που η κυρία Όουκεν έκανε την αναφορά που έκανε στο τέλος, γιατί αυτές οι αντιπροσωπείες οι οποίες ασχολούνται με πολύ ευαίσθητα θέματα, θα πρέπει να τύχουν μεγάλης προσοχής. Στην περίπτωση της Βουλγαρίας, ένας από τους συναδέλφους έφυγε τελευταία στιγμή και έγινε μια προσπάθεια να μην θεωρηθεί έτσι πολιτική δράση ή κίνηση κατά των σοσιαλιστών και είπαμε ότι πρέπει να υπάρχει και ένας από τους πράσινους επίσης. Πάντως, πάντως λέω, πρέπει να αποφύγουμε να εμπλεκόμαστε ε, σε εσωτερικές διαμάχες, γιατί αυτό τελικά θα αποβεί ε, προς ε, ζημίαν μας. Και βεβαίως εδώ παίζεται και το καλό όνομα της Επιτροπής μας, γιατί οι πολίτες στρέφονται στην Επιτροπή Αναφορών ε, σαν να είναι πραγματικά η τελευταία τους δυνατότητα προσφυγής. εάν διαπιστώσουν ότι κανείς δεν ενδιαφέρεται για αυτούς, ότι προσπαθεί να τους ε, χειραγωγήσουν, γιατί στην περίπτωση μας, στην περίπτωση που μας απασχολεί, ε, ένας από τους αναφέροντες ε, θεωρήθηκε persona non grata ε, και πραγματικά είχαμε και την αίσθηση ότι όλοι αυτοί οι άνθρωποι, οι αναφέροντες, ήταν παρείες που δεν μπορούσαν να μπουν στην αίθουσα και δεν μπορούσαν να μιλήσουν, απλώς γιατί ήθελαν να προστατέψουν τα όρη ρίλα. Αυτά είναι μερικά, αυτές είναι μερικές από τις ανησυχίες μας, ε, οι οποίες ε, δεν αποτελούν έτσι, μεροληπτικά σχόλια, ε, ούτε προσπαθώ να πάρω το μέρος του ενός ή του άλλου λέγοντας όσα είπα. Όμως είναι πάρα πολύ σημαντικό να επιστήρουμε την προσοχή των εθνικών κυβερνήσεων ότι είναι απαράδεκτος αυτός ο τρόπος δράσης. Δεν είναι δυνατόν να αντιτιθέμεθα στην ευρωπαϊκή πολιτική. Σας ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Θα ήθελα και εγώ με τη σειρά μου να ευχαριστήσω την κυρία Όκεν για την ιδιαίτερα επαγγελματική στάση που έδειξε η αντιπροσωπεία. Θα ήθελα επίση να την ευχαριστήσω για την παρουσίαση την οποία μόλι έκανε. Να ευχαριστήσω επίσης και τη γραμματεία της Επιτροπής Αναφορών για τη διοργάνωση της παρουσίας της αντιπροσωπείας της Επιτροπής Αναφορών Επιτόπου στην Βουλγαρία. Θα ήθελα λοιπόν να ευχαριστήσω όλους τους συμμετέχοντες. Όσον αφορά τα σημεία στα οποία αναφέρθηκαν οι συνάδελφοι, δεν θα ήθελα να επαναλάβω τα όσα είπαν, να επιμείνω σε δύο σημεία. Όσον αφορά τις γενικότερες συστάσεις για το πώς θα πρέπει να διοργανώνεται μια αντιπροσωπεία βάσει του παραδείγματος της Βουλγαρίας, ναι, συμφωνώ, θα ήθελα όμως να επιμείνω στο εξή σημείο. Για μένα το σημαντικότατο πρόβλημα το οποίο εντοπίσαμε επιτόπου είναι η απουσία διαλόγου ανάμεσα στις τοπικές αρχές και τους αναφέροντες. Το ζήτημα αυτό είναι ο βασικότατος παράγοντας ο οποίος ε, επηρέασε, αν θέλετε, τον τρόπο που εξελίχθηκε η αντιπροσωπεία και τις συζητήσεις που γίνανε. Δεν νομίζω ότι μπορούν να επιληθούν τα προβλήματα αν απουσιάζει ο διάλογο. Θα πρέπει και από τι δύο πλευρέ, τόσο αναφέροντε όσο και τοπικέ αρχέ, να έχουν το θάρρο και να λένε ότι όντω δεν ήρθαμε σε επαφή, δεν είχαμε τη δυνατότητα να συζητήσουμε και προσπαθούμε τελικά να επιλύσουμε ένα πρόβλημα μέσω του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Για παράδειγμα, οι αναφέροντες του Σουκοντόλ δεν ήρθαν σε επαφή με τον δήμαρχο της Σόφιας εδώ και 1,5 χρόνο, με αποτέλεσμα να μην γνωρίζει τελικά ποιο είναι το πρόβλημα. Υπάρχει λοιπόν μια απουσία διαλόγου ανάμεσα στους αναφέροντες που εμεί γνωρίζουμε και στις τοπικές αρχές και ερχόμαστε κατά αυτόν τον τρόπο στο πρόβλημα αυτό που έχουμε εντοπίσει σε πάρα πολλές συνεδριάσεις μας. το τρίτο αυτό τμήμα, αν θέλετε, οι τρίτοι συμμετέχοντες οι οποίοι πολύ συχνά αποτελούν αντικείμενο της α, συζήτησής μας είναι οι άνθρωποι αυτοί οι οποίοι έρχονται τελικά σε επαφή με τις τοπικές αρχές, οι διαμεσολαβητές κατά κάποιο τρόπο. Ουσιαστικά όμως και αυτό εξηγεί για ποιο λόγο οι περισσότερες περιπτώσεις είναι πολύπλοκες, για ποιο λόγο υπάρχει απουσία άμεσου διαλόγου και για ποιο λόγο δυσκολευόμαστε πάρα πολύ να βρούμε κάποιες λίστα στα προβλήματα τα οποία εξετάζουμε. Άκουσα ότι ορισμένοι επιχειρηματίες είναι διεφθαρμένοι. Δεν μπορώ να μην αντιδράσω, κυρία Άουκεν. Πιστεύω λοιπόν θα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί όταν κάνουμε τέτοιες καταγγελίες. Θα πρέπει να γίνει μια διαφοροποίηση ανάμεσα στην κατάσταση την οποία είδαμε επιτόπου και στις, στους κανόνες που ισχύουν για τις εταιρικέ σχέσεις δημοσίου-ιδιωτικού τομέα δεν θα πρέπει προφανώς να είναι μόνο οι δημόσιες αρχές οι οποίες ε, διαχειρίζονται ένα σχέδιο, θα πρέπει να συμμετέχουν και οι ιδιώτες, έτσι δεν είναι. Και από την άλλη δεν θα πρέπει να έχουμε μόνο μία επιχείρηση, γιατί καταλαβαίνετε ότι πολλές φορές ε, αυτό θα μπορούσε να οδηγήσει ακόμα και στην καταστροφή της φύσης. Είναι πολύ σημαντικό να υπάρχει όμως μια εταιρική σχέση ιδιωτικού δημοσίου τομέα προς ε, όφελος των πολιτών και για την προστασία του περιβάλλοντος. Θα ήθελα επίσης να αντιδράσω σε σχέση με δύο σημεία τα οποία ακούστηκαν όσον αφορά την έλλειψη διαφάνειας. Η κυρία Ούκεν μας είπε ότι θα πρέπει να συνεχιστούν οι προσπάθειες, να σε υπενθυμίσω ότι όσον αφορά το σύστημα διοδότησης, ο νυν υπουργό περιβάλλοντο είναι αυτό ο οποίο εγγενίασε το νέο σύστημα διοδότηση, το οποίο ισχύει εδώ και ένα χρόνο και νομίζω ότι θα πρέπει να ενθαρρύνουμε την απόφαση αυτή. Ο ίδιο ο Πρωθυπουργό δημόσια στο διαδίκτυο ανήρτησε όλη την διαδικασία αδειοδότησης. Πριν το 2009 η διαδικασία ήταν εντελώ αδιαφανής. Τώρα τα πράγματα έχουν αλλάξει. Όσον αφορά την δυνατότητα που έχει η κυβέρνηση για την νομιμοποίηση κάποιων καταστάσεων, να σας πω ότι στις περισσότερες περιπτώσεις ασχοληθήκαμε με αναφορές του 2006, του 2007, του 2008. Επομένω, με χαροποιεί το γεγονός ότι ε, τώρα η κοινωνία των πολιτών μέσω της διαδικασίας υποβολής αναφορών ουσιαστικά λένε ξεκάθαρα τι θέλουν και πολλές φορές αντιδρούν ενάντια στις αρχές. Το βλέπω θετικά. Καταλαβαίνετε ότι κάτι τέτοιο δεν γινόταν τόσο ανοιχτά στο παρελθόν. Έχει αλλάξει πλέον η κατάσταση και εγώ ερμηνεύω τα πράγματα ως εξή. Πιστεύουν αυτή τη στιγμή ότι κάποια πράγματα μπορούν να γίνουν διαφορετικά, βλέπουν ότι τα πράγματα έχουν αλλάξει και τολμούν να έρθουν σε επαφή με τις ε, τοπικές αρχές ανοιχτά. Και αυτό ακριβώ ουσιαστικά είδαμε όταν ερχόμασταν σε επαφή με του αναφέροντε. Βλέπουν ότι τα πράγματα κινούνται προ την σωστή κατεύθυνση και γι' αυτό το λόγο και αυτοί συμμετέχουν πιο ανοιχτά, πιο ενεργά και επιθυμούν να βρεθεί η καλύτερη δυνατή λύση. Όσον αφορά τα διάφορα σημεία στα οποία αναφερθήκατε, συμφωνώ με την άποψή σα. Όντω έγινε μια έρευνα επιτόπου και τα πράγματα μιλούν από μόνα του. Θα ήθελα απλώ να επανέλθω στα όσα αναφέρθηκε, στα όσα αναφέρθηκε ο κύριος Μποστινάρου, κάνοντας κάποιες γενικές παρατηρήσεις όσον αφορά την διαδικασία διοργάνωσης μιας διερευνητικής επίσκεψης, μιας fact-finding mission. Θα ήθελα να πω κάτι το οποίο με αφορά και κάπως προσωπικά και κάτι το οποίο θα ήθελα να εκφράσω σαν ανησυχία τελικά. Στις 18 Ιουνίου έστειλε ένα email το οποίο δημοσιεύτηκε στον βουλγαρικό τύπο και με κατήγγυλαν ότι ουσιαστικά προσπαθούσα να σαμποτάρω την επίσκεψη που γινόταν στη Χωματερή. Ο αναφέρον επίσης είπε συγκεκριμένα ότι προσπαθούσα εγώ να εμποδίσω την διεξαγωγή της α, επίσκεψης αυτής. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι ο αναφέρον αυτόν που με κατηγορεί σε καμία περίπτωση δεν ήρθε σε επαφή μαζί μου, σε καμία περίπτωση δεν μου μίλησε ανοιχτά. Δεν μπορώ να καταλάβω πώς το email μου αυτό έφτασε στα χέρια του τύπου και ανησυχώ κάπως για το επίπεδο εμπιστευτικότητας των ε, email μας. Ελπίζω ότι κάτι τέτοιο δεν θα επαναληφθεί στο μέλλον. Γιατί πιστεύω ότι κάτι τέτοιο τελικά επηρεάζει πάρα πολύ τις συνθήκες στις οποίες εργαζόμαστε και σίγουρα οι συνθήκες αυτές ήταν δύσκολες και η πιο άμεση επίπτωση τελικά ήταν ότι ε, χρησιμοποίησαν την καταγγελία αυτή τα, ο, μάλλον, τα μέσα μαζικής ενημέρωσης της Βουλγαρίας και ουσιαστικά δώσαν ένα πολύ έντονο πολιτικό χαρακτήρα στην επίσκεψή μας. Υπήρχε μάλιστα ένα άρθρο σε μια εφημερίδα η οποία έλεγε ότι είναι ένα συγκεκριμένο πολιτικό κόμμα το οποίο υποδέχεται την αντιπροσωπεία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και χάρη στην συμβολή του πολιτικού αυτού κόμματος μόνο γίνεται πραγματικότητα η επίσκεψη αυτή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Κάτι τέτοιο δεν θα ήθελα να επαναληφθεί στο μέλλον. Γιατί α, ε, ουσιαστικά αυτό το οποίο είδαμε είναι ότι τα μέσα μαζική ενημέρωση στη Βουλγαρία εξαιτία του γεγονότο αυτού είχαν διαμορφώσει ήδη μια άποψη όσον αφορά την επίσκεψή μα. Κάτι το οποίο θα πρέπει να συμβαίνει. Συμφωνώ επίση με τα όσα είπατε κύριε Μποστινάρου ότι ε, το πρόγραμμα το οποίο καταρτίζεται εκ των προτέρων θα πρέπει να τυχαίνει απόλυτου συμβασμού, δεν θα πρέπει να τροποποιείται Είδαμε επίσης ότι ε, κάποια πράγματα παρερμηνεύτηκαν εξαιτίας κάποιων ε, αλλαγών που είχαν γίνει. Θα ήθελα να έρθω ίσως στο πιο σημαντικότερο σημείο της παρεμβασής μου αυτή τη στιγμή όσον αφορά τη συμπεριφορά των ε, μελών, κυρίως των μελών εξοφίσιο επί τόπου. Πιστεύω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό τα μέλη αυτά να προσπαθούν να είναι όσο δυνατόν πιο συγκρατημένα στην συμμετοχή τους, προκειμένου να μην αναμοχλεύουν τα πάθη, ιδίως από πολιτικής πλευράς. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να βοηθούν την ομαλή διοργάνωση των συναντήσεων, των συζητήσεων και να μην κάνουν δηλώσεις στον τύπο ή να μην δίνουν ε, παρασκηνιακά κάποιες συνεντεύξεις. Το σημαντικότερο είναι να βοηθούν ουσιαστικά την συμμετοχή των βουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που προσπαθούν σε κάθε περίπτωση να προωθήσουν με αμεροληψία τα συμφέροντα των πολιτών. Ολοκληρώνω στο σημείο αυτό λέγοντας ότι είτε το θέλουμε είτε όχι οι αποστολές ε, της Επιτροπής, της δικής μας Επιστροπής των Αφορών βρίσκονται πάρα πολύ κοντά στον πολίτη, ουσιαστικά ενσαρκώνουν την ε, σύνδεση αυτή, την άμεση που έχουμε με τον Ευρωπαίο πολίτη. Είναι πάρα πολύ σημαντικό πάντως για μας τους Ευρωβουλευτές να παραμένουμε αμερόληπτοι, αντικειμενικοί, να μην υποτασσόμαστε σε εθνικά πολιτικά συμφέροντα σε καμία περίπτωση θα πρέπει να αποτελούμε θύματα χειραγώγησης, γιατί καταλαβαίνετε ότι αυτό δημιουργεί τελικά αντιευρωπαϊκά συναισθήματα στον Ευρωπαίο πολίτη και αυτό το είδαμε στην ναζαρεη Μπαζαμπάνια. Θεωρώ ότι είναι τρομακτικό αυτό το ότι κάποιοι πολίτες είπαν ότι εμείς υποστηρίζουμε την Ευρώπη και αυτό το οποίο βλέπουμε είναι ότι η Ευρώπη δεν μας υποστηρίζει όμως καταλαβαίνετε ότι τέτοια παραδείγματα τελικά πυροδοτούν όλη αυτή την ε, αντιευρωπαϊκή ευρωσκεπτιστική στάση που βλέπουμε σε ορισμένου Ευρωπαίους πολίτες. Καταλαβαίνετε ότι σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει να χάνουμε την αξιοπιστία μας. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να βλέπουμε τις αρνητικές επιπτώσει ε, των ε, περιπτώσεων αυτών. Ας αντλήσουμε κάποια διδάγματα λοιπόν από τις αρνητικές αυτές εμπειρίες και Όπω είπα στην κυρία Όκεν και στον κύριο Μποστινάρου, είναι πάρα πολύ σημαντικό να καταλήξουμε σε κάποια θετικά συμπεράσματα από την αποστολή αυτή. Ευχαριστώ πολύ, αγαπητοί συνάδελφοι. Ε, συνάδελφε. Και βεβαίως σημειώνω τον προβληματισμό όσον αφορά την μεθοδολογία ε, που εφαρμόζεται στις επισκέψεις ε, και πραγματικά στο μέλλον θα πρέπει να το προσέξουμε. Είναι προφανές αυτό που ε, καταγγείλατε. Και ε, αυτό που συνέβη στη Βουλγαρία και μετά για τη Ρουμανία το έχουμε διαπιστώσει επανειλημμένα. Νομίζω ότι όλοι θα πρέπει θα πρέπει να γνωρίζουμε όλοι ότι η Επιτροπή μας είναι Επιτροπή για τους πολίτες, η οποία δεν θα πρέπει να πολιτικοποιείται, γιατί διαφορετικά εγχειρηματοποιείται ε, και χρησιμοποιείται λοιπόν από τα διάφορα εμπλεκόμενα μέρη ε, προς τη μία ή την άλλη κατεύθυνση. Επομένως θα πρέπει λίγο να αναθεωρήσουμε τις απόψεις μας, ώστε τέτοιου είδους στάσεις να μην διαπιστωθούν στο μέλλον. Όλα τα στοιχεία αυτά ε, βεβαίως ε, θα, ε, θα πρέπει να μας απασχολήσουν στο μέλλον. Πάντως, και κάποια ενδιαφερόμενα μέρη οπωσδήποτε θα πρέπει να συμμετέχουν σε τέτοιες αποστολές γιατί γνωρίζουν καλά και την κατάσταση. Θα δώσω το λόγο στην κυρία Ούκεν αλλά παρακαλώ πολύ έχουμε χάσει πολύ χρόνο και κάπως πρέπει να κερδίσουμε τον χρόνο. Έχουμε αναφέροντες εδώ. Θα ήθελα ευχαριστήσω τη Μαριάννα, αλλά πρέπει να τονίσω ξανά ότι πολλά μέλη, πολλά επίσημα στελέχη είναι πολύ εξυπηρετικά και φιλικά και πάντοτε βεβαίως αντιμετωπίζουμε διαφορές και διαμάχες μέσα στο πλαίσιο της πολιτικής γιατί η πολιτική πολλές φορές είναι και βρώμικη υπόθεση. Ε, πιστεύω λοιπόν ότι δεν θα δεν θα έλεγα ότι πρέπει να προσπαθήσουμε να σβήσουμε, να διαγράψουμε, να ξεφορτωθούμε όλες αυτές τις πολιτικές διαφορές, γιατί αυτό δεν το καταφέρουμε ποτέ. Οι πολιτικές διαφορές και διαμάχες είναι μέρος της πολιτικής ζωής. Ευχαριστώ λοιπόν όλους ξανά και ιδίω τη Γραμματεία για τις προσπάθειές της. Η οργάνωση ήταν εξαιρετική πρέπει να αναγνωρίζουμε ποιος κάνει αυτή την καταπληκτική εργασία. Ευχαριστώ. Ο Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Μια σύντομη προσθήκη επί της διαδικασίας. Δεν μπορούμε να κλείσουμε το στόμα κανενός ε, βουλευτή ή πολιτικού αυτό ισχύει και για την άλλη πλευρά αλλά και για μας, για τα μέλη της αντιπροσωπείας. Σε αυτά τα ταξίδια και στην προετοιμασία των ταξιδιών ε, μας είχαν πει ότι οι βουλευτές του κράτους φιλοξενίας, ας πούμε, του κράτους υποδοχής, ε, μπορούν να μας δώσουν χρήσιμες συμβουλές και στοιχεία, ε, παρόλο που μπορεί να μην είναι επίσημα μέλη της ε, αντιπροσωπείας λοιπόν, πιστεύω ότι είναι άδικο να εμποδίζονται αυτοί οι άνθρωποι να μπορούν να έρθουν σε επαφή μαζί μας για να μας δώσουν πληροφορίες, ας πούμε, και χρήσιμες οδηγίες κλπ. Ελπίζω να μην ξανασυμβεί αυτό ε, και το ξαναλέω, εμείς είμαστε Επιτροπή Αναφορών, είμαστε εκεί για τους πολίτες, η δουλειά μας είναι για τους πολίτες και όχι για να εκμεταλλευτούμε την κατάσταση για προεκλογικές εκστρατείες, καμπάνια προβολή κλπ. Επίσης, ε, ευχαριστώ ε, που δεν είχε, ε, πρέπει να είμαστε ευγνώμενες που δεν αποσύρθηκε λόγω της προσβολής που της έγινε, αλλά προσπάθησε να διευκρινίσει την κατάσταση και ευχαριστώ πάρα πολύ τη συνάδελφο για αυτήν την στάση, τη μεγαλοψυχία της. Ο κύριος Ταλευράς. From Bulgaria, <clears throat> Uh, the Θα uh, ευχαριστώ πάρα πολύ ε, την ενημέρωση αυτή που μας έγινε για τις δύο επισκέψεις. Ε, πολλά αναφέρθηκα στον τύπο και δύο πράγματα τα οποία μου έκαναν εντύπωση. Το ένα είναι ότι οι πολίτες πρέπει να να συμμετάσχουν περισσότερο στις εργασίες. Τους ενδιαφέρει και για μια ευρύτερη συμμετοχή ε, και πολλές φορές δεν υπάρχει αυτός ο χρόνος. Δεν εννοώ τους αναφέρονται συγκεκριμένα, αλλά γενικά ομάδες ε, των, του πληθυσμού, των κατοίκων, οι άνθρωποι. Λοιπόν, ευρύτερη συμμετοχή του κοινού. Δεύτερον, ε, αυτή η κατάσταση δεν είναι πρόσφατη, είναι ε, ε, ε, κρίσιμη εδώ και 5-6 χρόνια. όχι μόνο όσον αφορά τις αναφορές, αλλά έχει επιπτώσεις σε όλο τον πλησισμό, που προσπάθησε να εξηγήσει τι συμβαίνει τέλος πάντων. Πώς εξηγείται αυτή η κατάσταση. Πάρα πολλοί πολίτες ανησυχούν δεν θα επισκεφτήκατε, πιστεύω, ε, την ε, τοποθεσία συσκευασία των απορριμμάτων, όπου πακετάρονται τα απορρίμματα. Ένα μεγάλο μέρος αυτών των απορριμμάτων βρίσκεται ακόμα στη χωματερή που βρωμάει ε, ε, συνεχεία μεταφέρονται και ε, εναποθέτονται παντού στη Βουλγαρία, πάνω από εδώ, πάνω από εκεί και αναρωτιούνται οι πολίτες τι γίνεται. Δεν αφιβάλλω ότι, έχετε τη σωστή, ότι υπάρχει σωστή προσέγγιση εκεί, αλλά η απόθεση και διαχείριση απορριμμάτων της πρωτεύουσα της Σόφιας είναι ένα πρόβλημα που καίει τους κατοίκους και σας χαίρω που κάνετε αυτή την εξαιρετική ε, εργασία με την επίσκεψή σας, διότι επικεντρήξατε τον προ, τους προβολείς πάνω στο θέμα. Ευχαριστώ. Ο κύριος Μπρέκλαντ από την Επιτροπή. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Θα μιλήσω κι εγώ για μία φορά στη δική μου μητρική γλώσσα όπως έκανε η κυρία Όκεν. Μερικές τεχνικές παρατηρήσεις. Βεβαίως καταλαβαίνουμε όλοι ότι πρόκειται για ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα Ενδεχομένως καλό θα ήταν να αναφέρομαι ότι ε, την 1η Ιουλίου η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε ε, το πρώτο ε, τμήμα 40 εκατομμύρια ευρώ για τρία χρόνια έτσι ώστε σιγά σιγά να λυθεί το πρόβλημα αυτό. Ενεκρίθη λοιπόν αυτό το πρώτο τμήμα της χρηματοδότησης. Προς τον κύριο Μποστινάρου να πω ότι δεν πιστεύουμε με μεγάλη αφέλεια όλα όσα μας σερβίρουν ή μας λένε οι τοπικές αρχές. Ε, βεβαίως ερχόμαστε σε επαφή και με τους αναφέροντες ε, ε, και γι' αυτό ακριβώς ξεκινούμε διαδικασίες επί για περιπτώσει όπω αυτή η χωματερή ή και άλλε. Θα δείτε και το Σεπτέμβριο ότι θα υπάρξουν πολλέ διαδικασίε επί παραβάση. Απ' την άλλη πλευρά έχετε απόλυτο δίκιο διότι καταδεικνύεται μία ε, έλλειψη του συστήματος ε, για την ώρα όσον αφορά τα περιβαλλοντικά ζητήματα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν έχει δικαίωμα επιθεώρηση, αλλά ξέρετε ότι έχουμε μία διάσκεψη, την είχαμε μάλλον τη 15η Ιουνίου ε, που μα έκαναν την τιμή να συμμετάσχουμε συμμετάσχουν και η κυρία Ούκεν και η Πρόεδρος ε, ε, και βεβαίως αυτό είναι το κυριότερο ζήτημα για μας, ε, δηλαδή η δυνατότητα επιθεώρησης που θα πρέπει να δοθεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέσω κάποιας υπηρεσίας. Εδώ έχουμε μεγάλο πρόβλημα λοιπόν, δεν μπορούμε επιτόπου να συλλέξουμε αποδεκτικά στοιχεία. Περιμένουμε τους αναφέροντες, περιμένουμε εσάς, περιμένουμε τους καταγγέλλοντες να μας δώσουν συγκεκριμένα στοιχεία. Αυτό είναι όντως ένα ζήτημα πολιτικό. Ευχαριστώ πολύ και ευχαριστούμε και για τη συνεργασία σας. Νομίζω ότι είναι ένα άνοιγμα το οποίο μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε και στο μέλλον, λέει η Πρόεδρος. Νομίζω ότι μπορούμε να ολοκληρώσουμε τη συζήτηση του σημείου αυτού. Θα επανέλθουμε βεβαίως όταν θα υποβληθεί η έκθεση. Σημείο 13, ε, αναφορά 1026 του 2010 του Ράντο στην Ρούσε, βουλγαρικής ηθαγένειας, ο κύριος Στάντσεφ εξ ονόματος του υπογράφοντος. Δίνω το λόγο λοιπόν στον κύριο Στάντσεφ για πέντε λεπτά. Уважаеми дами и господа евродепутати, казвам се Валери Станчев и се явявам пред вас в качеството си на представител на господин Радостин Русев, за да изложа резюме на петицията, подадена от него, касаеща злоупотреби и корупция в България и в частност град Сливен υπάρχει ένα, πολιτικό, ε, συγγνώμη, ένα τεχνικό ζήτημα από ό,τι φαίνεται. Ε, Πρόκειται, η αναφορά αυτή ε, επικεντρώνεται στη διαφθορά στη Βουλγαρία. Δεν μπόρεσε να έρθει ο αναφέρον διότι είναι, σε μια, είναι στο δικαστήριο διότι η δίκη ορίστηκε για σήμερα. ο δήμαρχος του Σλίβεν και οι τοπικοί άρχοντες εκεί της ε, περιφέρειας του έχουν καταχραστεί ε, πόρους, έχουν, υπάρχουν μεγάλες ατασταλίες ε, στο Δήμο αυτό. Η ΙΣΠΑ έδωσε κονδύλια για το σύστημα αποχέτευσης και ίδρυυσης και το έργο το ανέλαβε η εταιρεία Hydro Systems σε βάση της διαδικασίας δημοσίων ε, συμβάσεων. Όμως ε, το έργο αυτό το σταμάτησε παράνομα ο Δήμαρχος, εν συνεχεία βεβαίως ε, σημειώθηκε καθυστέρηση του έργου και εν συνεχεία σταμάτησε. Η δικαιολογία του Δημάρχου για να σταματήσει το έργο ήταν ότι η εταιρεία Hydro Spa αρνήθηκε να χρησιμοποιήσει έναν υπεργολάβο ο οποίος ήταν, φίλος του Δημάρχου. Αρνήθηκε λοιπόν η εταιρεία αυτή στην οποία ανατέθηκε το έργο με κονδύλια της Ευρωπαϊκής Ένωσης να χρησιμοποιήσει ε, ε, μια εταιρεία υπεργολαβική που ήταν φίλη προσκύμενη προς τον Δήμαρχο. Επίσης, ε, συνεχεία, η ανα οι επισκευές ενός οίκου ευγυρίας στο Σλίβεν και εκεί σημειώθηκαν οι ε, οικονομικές ατασταλίες και παρόμοιες ατασταλίες σημειώθηκαν επίσης στην επισκευή του συστήματος ίδρευσης του, στις διάφορες περιοχές του Σλίβεν. Ε, όπως επίσης τα δημόσια λουτρά και σε διάφορες γειτονιές του Σλίβεν. Η εταιρεία Poolgate είχε αναλάβει το έργο, εν συνεχεία όμως πήγε στα χέρια εταιριών και υπεργολάβων φιλικών πάλι προς το Δήμαρχο. Οι ατασταλίες αυτές λοιπόν και παρανομίες αναφέρονται σε ε, χειραγώγηση των συμβάσεων, 177 εκατομμύρια λεβ είναι η, το ύψος των αναθέσεων αυτών και λόγω των παράνομων αναθέσεων και ατασταλιών που σημειώθηκαν δεν θα μπορέσουμε να προσελκύσουμε άλλες ε, ευρωπαϊκές, ε, ευρωπαϊκές πιστώσεις αρμόδια αντιδήμαρχος ήταν και λογίστρια της περιφέρειας Κλίτσκοφ και αυτή τη στιγμή είναι υπεύθυνη, υπεύθυνη με τον Δήμαρχο για αυτές τις παρανομίες. Μία άλλη εταιρεία και πάλι ήταν υπεύθυνη για παράνομες ε, οικονομικές ενέργειες σε μια άλλη περιφέρεια της Βουλγαρίας και εμπλέκεται και αυτή στην περιοχή του Σλίβεν λόγω του Δημάρχου. Και δεδομένου ότι όλα αυτά τα έργα ή έχουν σταματήσει ή δεν συνεχίζονται ή έχουν γίνει με ε, κακό τρόπο και δεν καλύπτουν τις ανάγκες του τοπικού πληθυσμού. Οι κάτοικοι έχουν αγανακτήσει, 24 ε, κάτοικοι υπέγραψαν ένα αίτημα διαμαρτυρίας, όμως δεν ακούστηκε η φωνή τους καθόλου. Ε, άλλα έργα έχουν απορροφήσει 3,5 εκατομμύρια γιούρος υπό την αιγίδα της ΙΣΠΑ βεβαίως, υποτίθεται για τεχνική βοήθεια άλλα κονδύλια δηλαδή τα οποία έχουν χαθεί και ο ανάδοχος ήταν η εταιρεία Aquaculture 25.000 ε, ευρώ απορροφήθηκαν χωρίς να υπάρχει δημόσια διαδικασία και δημόσια ανάθεση, απλώς ε, πήγαν από τσέπη σε τσέπη τα χρήματα. Και πάλι ο δήμαρχος Λέτσκοφ είναι σαφώς υπεύθυνο για αυτή την ε, ατασταλία, ε, γιατί είναι υπεύθυνο για τη διαχείριση των κονδυλίων από την ΙΣΠΑ. Μία άλλη ε, εταιρεία Club Economic 2000 διαχειρίζεται προγράμματα εκατομμυρίων ευρώ ε, και σε όλες αυτές τις αναθέσεις ε, βλέπουμε ότι έχει παραβιαστεί διαδικασία δημόσιας ανάθεσης, δημοσίων συμβάσεων, υπεργολαβιών κλπ. Και τα έχουν οδηγήσει στη χρεοκοπία επιχειρήσεων, σε ανεργία και στην, η όλη αυτή κακοδιαχείριση ε, οφείλεται ε, στην κατάχρηση εξουσίας του Δήμαρχου και του τοπικών αρχών το δικαστήριο έχει αρνηθεί να ακούσει ε, τις ε, κατηγορίες αυτές. Ε, εκκρεμούν τέσσερις ποινικέ διαδικασίες ενώπιον των δικαστηρίων. Ο Υπουργός Εσωτερικών και άλλες υψηλότερες πολιτικές αρχές έχουν δείξει μέσα στον τύπο και στα ηλεκτρονικά μέσα ότι προστατεύουν και καλύπτουν αυτή τη διαφορά. Θέλουμε λοιπόν να υπάρξει μία αξιολόγηση και μία έρευνα της κατάστασης αυτής από ανεξάρτητα θεσμικά όργανα. Κυρίες και κύριοι και εκ μέρους του ετούντος κυρίου Ρούσεφ θα ήθελα να σας ευχαριστήσω που με ακούσατε και για την προσοχή που δώσατε σε αυτή την υπόθεση. Πιστεύουμε στην ε, δύναμη του νόμου και στην ευρωπαϊκή νομοθεσία. Πιστεύουμε ότι η Βουλγαρία θα μπορέσει με τη βοήθειά σας να ακολουθήσει ε, τον ίδιο δρόμο όπως τα άλλα κράτη-μέλη. Ο δρόμος αυτός πρέπει να είναι αδιάβλητος και να μην σημειώνονται ατασταλίες και, δια... και δια... Ε, περιπτώσεις διαφθοράς. Ευχαριστώ, λέει η πρόεδρος, δίνω το λόγο στην ε, Κομισιόν. Καλημέρα σας. Τα έργα αυτά απαρτίζονται από δύο τμήματα ουσιαστικά. Θα ήθελα να σας εξηγήσω πώς εμπλεκόμαστε εμείς από τη Γενική Διεύθυνση Περιφερειακής Ανάπτυξης. Το 2010, κατά τη διάρκεια μιας αξιολόγησης που κάναμε στα πλαίσια του σχεδίου ΙΣΠΑ, ότι η πολιτεία εκεί χρησιμοποιούσε κάποιες συμβάσεις πλαίσιο για την κατασκευή, για την οικοδόμηση κάποιων κτηρίων. Συμβάσεις πλαίσιο τέτοιες χρησιμοποιούνται αρκετά σπάνια. Εμείς εκφράσαμε την αντίρρησή μας ως Ευρωπαϊκή Επιτροπή και σε μια περαιτέρω αξιολόγηση που κάναμε ζητήσαμε να μας δοθούν περαιτέρω πληροφορίες όσον αφορά τη συγκεκριμένη αυτή σύμβαση, αυτές τις συμβάσεις πλαίσιο. Στείλαμε όλες τις πληροφορίες στην DigiMart, αξιολόγησαν τις πληροφορίες αυτές, το όλο πακέτο μέτρων και στις 22 Ιουνίου λάβαμε ένα έγγραφο στο οποίο λέγεται ξεκάθαρα ότι αυτές οι ε, συμβάσεις πλαίσιο δεν συνάδουν με τις αρχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις δημόσιες συμβάσεις και ότι υπήρχε και μία περίπτωση στρέβλωσης του ανταγωνισμού η οποία δικαιολογείται βάσει συγκεκριμένων ευρημάτων. Στις 26 Ιουνίου στη συνέχεια η Ευρωπαϊκή Επιτροπή απέστειλε μία επιστολή προς τον Υφυπουργό Περιβάλλοντος στην οποία εξηγούσε ότι ακριβώς επειδή δεν είχε ακολουθηθεί η ε, σωστή διαδικασία για αυτές τις δημόσιες συμβάσεις, έπρεπε να επιβληθούν κάποια μέτρα και ότι ως Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν θα παρατείναμε το σχέδιο ΙΣΠΑ για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. και ουσιαστικά το σχέδιο αυτό συνδέεται και με άλλα σχέδια περιφερειακής ανάπτυξης στη χώρα. Αυτή λοιπόν την εβδομάδα, πριν το τέλος της ε, τρέχουσας εβδομάδας, θα στείλουμε ένα οριζόν, μια οριζόντια επιστολή στον Υπουργό Ντόνισεν, ζητώντας του να εξασφαλίσει ότι τουλάχιστον στο μέλλον όλες αυτές οι ε, δημόσιες συμβάσεις πλαίσιο θα διεξάγονται με πολύ προσεκτικό τρόπο και ότι θα αποφεύγεται κάθε περίπτωση αγωνισμού. Αυτά όσον αφορά την πλευρά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και όσον αφορά την αξιολόγηση την οποία κάναμε. Ελπίζω ότι θα λάβουμε κάποιες πληροφορίες για τις άλλες πλευρές των συμβάσεων αυτών. Ευχαριστώ πολύ, λέει η Πρόεδρος. Θέλει κανείς να πάρει το λόγο, ο πιο... Αυτό που μας παρουσίασε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην ουσία επιβεβαιώνει ότι σε αυτή την περίπτωση έχουμε πρόβλημα. Αυτό είναι το πρώτο στοιχείο. Εάν υπάρχουν προβλήματα, τα προβλήματα πρέπει να αντιμετωπιστούν. Και μπορούμε να το κάνουμε αυτό σε δύο επίπεδα. Το ένα είναι το βουλγαρικό, από το τοπικό επίπεδο μέχρι το κυβερνητικό και το άλλο είναι το επίπεδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και εδώ δεν άκουσα τίποτα ακόμα για την αντίθεση συμφερόντων, τη σύγκρουση συμφερόντων, εάν, υπάρχουν, εάν υπάρχει σύγκρουση συμφερόντων στην, που εμποδίζει την έρευνα της υπόθεσης. Εάν υπάρχει σύγκρουση συμφερόντων θα πρέπει να έχει το λόγο η Όλαφ, το Όλαφ. Και το Όλαφ, ο ρόλος του Όλαφ είναι πάρα πολύ δύσκολος όταν εμπλέκονται κοινοτικά, η κονδύλια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι δύσκολο να δράσει γρήγορα και αποτελεσματικά. Η ερώτησή μου είναι, τι θα γίνει εάν στο τέλος της ημέρας <laughs> έχετε την, τις αποδείξεις ότι οι ατασταλίες και η διαφθορά, η οποία βεβαίως είναι εις βάρος των πολιτών του Σλίβεν, τι θα γίνει λοιπόν με αυτή την περίπτωση και εσείς προσπαθήσετε να πιέσετε τη βουλγαρική κυβέρνηση να πάρει αποφάσεις επιτέλους. Πιστεύω ότι πρέπει να ασκηθεί αυτή η πίεση. Διότι η εικόνα του Σλίβεν σήμερα είναι εικόνα ενός ε, βομβαρδισμένου τοπίου μετά από πόλεμο, διαδομένου ότι υπάρχουν ερήπια παντού, ε, δεν έχουν ε, ολοκληρωθεί τα έργα, ημιτελή έργα, κτίρια και εγκαταστάσεις, η υποδομή λοιπόν είναι ημιτελής και άχρηστη και θα έλεγα η, προτείνω η αναφορά αυτή να παραμείνει εκρεμή πριν, έως ότου λάβουμε διευκρινήσεις από τη βουλγαρική πλευρά και την πλευρά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και περιμένω ε, μια πλήρη έκθεση των ατασταλιών ε, στην διαχείριση των ευρωπαϊκών πιστώσεων. Η κυρία Τσέρα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Και εγώ πιστεύω ότι αυτή η αναφορά πρέπει να παραμείνει ανοιχτή μέχρι ότου έχουμε όλες τις απαραίτητες πληροφορίες στα δύο επίπεδα ε, και από τις βουλγαρικές αρχές και από την Κομισιόν για να μπορέσουμε να διαμορφώσουμε τη θέση μας. Πιστεύω ότι αυτή η αναφορά περιλαμβάνει ε, διάφορα στοιχεία που πρέπει να ληφθούν σοβαρά υπόψη. Καταρχάς, Είμαι πολύ ευτυχής που άκουσα από την Κομισιόν ότι θα εξακολουθούν να συλλέγουν και να μας ενημερώνουν για τις πληροφορίες και τις διαδικασίες που εφαρμόζει η Όλαβ έτσι ώστε να έχουμε αξιόπιστες πληροφορίες από πλευράς Κομισιόν και Όλαβ. Από την άλλη πλευρά ε, πρέπει να λάβουμε και όλες τις απαραίτητες πληροφορίες από τις νόμιμες αρχές ε, της Βουλγαρίας έχουν γίνει επιθεωρήσεις έλεγχοι από τις αρμόδιες ελεγκτικές αρχές και ποια είναι τα αποτελέσματα Το δεύτερο θέμα που μπορούμε να εξετάσουμε είναι η εφαρμογή της νομοθεσίας δημοσίων συμβάσεων, η οποία συντάχθηκε με τη βοήθεια και την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι αρμόδια η οδηγία 17 για τις δημόσιες συμβάσεις. Πώς έχει εναρμονιστεί η κοινοτική νομοθεσία. Το βασικό πρόβλημα από ό,τι καταλαβαίνω είναι η σύμβαση πλαίσιο ε, υπό την ομοθεσία δημοσίων συμβάσεων στη Βουλγαρία. Υπάρχει και ένα άλλο έντυπο, υπάρχει και μια άλλη δομή που αποκαλείται ε, πλαίσιο συμφωνία. Συμφωνία πλαίσιο ή σύμβαση πλαίσιο. Θέλω να ξέρω εάν αυτές, αυτή η διαφορετική ορολογία σημαίνει και διαφορά στη φύση των συμβάσεων και στις υποχρέωσεις. Ε, Πρέπει και συμφωνώ με όλους τους προλαλήσαντες να περιμένουμε μέχρι ότου συλλέξουμε όλα τα απαραίτητα στοιχεία ώστε να μπορέσουμε να διαμορφώσουμε μία ουδέτερη και αντικειμενική γνώμη και να βρούμε τη σωστή λύση και να απαντήσουμε σωστά στον ετούντα. Ευχαριστώ συνάδελφε Νιντελτζέβα. Η κυρία Νιντελτζέβα υπέβαλε ερωτήματα τα οποία η αναφέρουσα ενδεχομένως μπορεί να απαντήσει. και να δούμε αν υπάρχει δυνατότητα να ε, προσκομιστούν επιπλέον στοιχεία τεκμηρίωσης, μια και ε, υπάρχει συγκεκριμένο αίτημα όσον αφορά την προέλευση των στοιχείων. Ε, καλό θα ήταν λοιπόν να αποσαφινιστούν περαιτέρω τα στοιχεία αυτά και ενδεχομένως να έχουμε ένα γραπτό, κάτι γραπτό. Επί της αναφοράς αυτής Βεβαίως ε, θα πρέπει να παραμείνει ανοιχτή η συζήτηση γιατί και η Επιτροπή και η Όλαφ... Α, συγγνώμη, θέλει κάποιος να πάρει το λόγο. Ε, ε, κύριοι συνάδελφοι, παρακαλώ πάρα πολύ να ζητάτε το λόγο ε, εξ αρχής, ε, έτσι ώστε να μπορώ να ρυθμίσω τη συζήτηση να ξέρω πόσοι θέλουν να βάλουν τον λόγο. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Θα ήθελα να κάνω κάποιες παρατηρήσεις. Εξαιτία του ζητήματο αυτού αποφάσισα να έρθω και εγώ σήμερα εδώ και να συμμετέχω στη συζήτηση. Ξέρετε ότι υπάρχει ένα ολόκληρο ιστορικό στην υπόθεση αυτή. Γνωρίζουμε ότι το πρόβλημα αυτό εφίσταται εδώ και 1,5 χρόνο. Από προσωπική πλευρά πρέπει να σα πω ότι έλαβα πάρα πολλά παράνο, παράπονα και καταγγελίε, γιατί όπω είπε ο κύριο Μποστινάρου, στην πόλη του Σλίβεν η εικόνα είναι η εικόνα ενός βομβαρδισμένου τοπίου. Εδώ και 1,5 χρόνο η κατάσταση δεν έχει αλλάξει. Το κέντρο, οι βασικοί δρόμοι της πόλης αυτής δεν είναι προσβάσιμοι. Καταλαβαίνετε τα σημαντικότα προβλήματα, τα προβλήματα που αντιμετωπίσουν οι πολίτες που κατοικούν στην περιοχή. Επισκέφθηκα λοιπόν την πόλη του Σλίβεν πέρυσι και είδα κι εγώ η διεισόμαση τι πραγματικά γίνεται, αφού είχε λάβει και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κάποιε πληροφορίε. Ήταν αδύνατο να καταφέρει να μετακινηθεί κανεί στην πόλη αυτή με το αυτοκίνητο. Και έστειλα μία επιστολή στον, στην, στον Υπουργό Ντόλτσεφ και από ό,τι άκουσα και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα αποστείλει μία επιστολή στον Υπουργό αυτό. Μα εγώ το έκανα πριν από πολύ καιρό και δεν κατάφερα τελικά να λάβω μία απάντηση και δεν το έκανα από πολιτικό συμφέρον. Ουσιαστικά προσπαθούσα να εκφράσω τα παράπονα των πολιτών και από ό,τι κατάλαβα υπάρχουν και πολλά κοινοτικά κονδύλια τα οποία έχουν δοθεί στην πόλη αυτή. Η απάντηση που μου έδωσε λοιπόν ο Υπουργό Ντόλτσεφ, ο οποίο είναι επικεφαλή για τα ευρωπαϊκά αυτά προγράμματα στη Βουλγαρία, ήταν. Τι να σας πω, μπορώ να σα στείλω μια επιστολή. Δεν έλεγε τίποτα απολύτως η επιστολή του αυτή δηλαδή δεν είχε κανένα ουσιαστικά περιεχόμενο η απάντησή του. Πράγμα το οποίο καταδεικνύει ότι σε ύψιστο επίπεδο στην βουλγαρική πολιτική γίνεται μία απόπειρα συγκάλυψης. Ακόμη και σήμερα τα πράγματα παραμένουν απαράλλαχτα. Τα πάντα έχουν σταματήσει εδώ και δύο σχεδόν χρόνια. Το ερώτημα λοιπόν το οποίο απευθύνω στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι το ακόλουθο. Στην επιστολή προς εσάς της 3ης Μαρτίου λένε ότι ακόμα περιμένουν να λάβουν την πλήρη τεκμηρίωση όσον αφορά τη σύμβαση πλαίσιο. Αν λάβετε υπόψη σας πώς ζουν οι 100.000 πολίτες της πόλης αυτής εδώ και δύο χρόνια που βιώνουν καθημερινά την κατάσταση αυτή, νομίζω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να ανησυχήσει λίγο περισσότερο καμία απολύτω βελτίωση δεν έχει επέλθει. Η, αυτή, αντιληγή αυτή επίσημων επιστολών ουσιαστικά δεν συμβάλλει σε τίποτα αυτή τη στιγμή. Πρέπει να τονίσω πώ είναι η κατάσταση. Ξέρω ότι υπάρχουν προβλήματα, ιδίω στο Υπουργείο Περιβάλλοντο τη Βουλγαρία. Μολονότι, ότι, όπω σα είπα, η προστασία και η συγκάλυψη γίνεται σε ύψιστο επίπεδο. Πώ θα επιλύσετε όμω την κατάσταση. Εδώ και δύο χρόνια οι Ευρωπαίοι πολίτε τη πόλη αυτή υποφέρουν εξαιτία τη κατάσταση. Για ποιο λόγο να μην πάτε, αν μη τι άλλο, να επισκεφτείτε την πόλη αυτή, να δείτε κι εσείς πώς έχει η κατάσταση. Φοβάμαι ότι αν διονυστεί το πρόβλημα αυτό, θα λάβουμε και άλλα παράπονα και άλλες καταγγελίες. Νομίζω ότι ε, τα δύο χρόνια αρκούν ακόμα και για την Όλαφ. Πρέπει να ξέρουμε πώς έχει η κατάσταση. Δεν τάσσομαι ούτε με τη μία, ούτε με την άλλη πλευρά. Πρέπει όμως να δούμε πού πρέπει να επικεντρωθεί η ευρωπαϊκή δράση είναι σαφέ ότι σε εθνικό επίπεδο δεν δίνονται απαντήσει αυτή τη στιγμή. Κάτι πρέπει να κάνει η Ευρώπη. Ευχαριστώ. Ε, Ευχαριστώ πολύ για αυτά τα σημαντικά στοιχεία που προσθέσατε. Και βεβαίως ε, ίσως ζητήσουμε και από την Όλαφ ε, να επιταχύνει λίγο την διερεύνηση του θέματος που αποτελεί αντικείμενο της αναφοράς. Και πάντως απαντούμε στον αναφέροντα ότι αφήνουμε ανοιχτό το ζήτημα της αναφοράς. Θα περάσουμε τώρα στο επόμενο σημείο. Αίτηση, αναφορά συγγνώμη του κύριου Τσιπριάν Ντόμπρε, Ρουμανική Ιθαγένεια, σχετικά με προβλήματα που προκύπτουν από την χρησιμοποίηση και διαχείριση από τη Ρουμανική κυβέρνηση των πιστώσεων του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου αγροτικής ανάπτυξης. Εδώ ε, καταδεικνύεται ότι δεν έχουν γίνει, δεν έχουν ακολουθηθεί σωστά οι διαδικασίες όσον αφορά ε, την πλήρωση των προϋποθέσεων ε, και των όρων του διαγωνισμού. Δεν είναι εδώ ο αναφέρον. Ε, πάντως ε, έχουμε συγκεκριμένα στοιχεία σχετικά με τον τρόπο καταμέτρησης ε, κάποιων πόντων που προϋπέθεται ο διαγωνισμός. Θα δώσω το λόγο στον κύριο Παπαδημητρίου. thank you. Κυρία Παπαδημητρίου, συγγνώμη. Since uh, the petitioner is not here, I will try to make a very brief resume on his uh, uh,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 Παρακαλώ ακούτε την ελληνική διερμηνία διότι είχα ένα τεχνικό πρόβλημα με το μικρόφωνο. Αν ακούτε την ελληνική διερμηνία καλά μπορείτε να κάνετε ένα διακριτικό νεύμα παρακαλώ στην καμπίνα 7. 7. Μας ακούτε παρακαλώ στην καμπίνα 7. Μπορείτε να κάνετε ένα διακριτικό νεύμα. Αν μας ακούτε στην καμπίνα 7. Μας ακούτε παρακαλώ στην καμπίνα 7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 Παρακαλώ, ακούγεται ελληνική διερμηνία από την καμπίνα 7. Μπορείτε να μας κάνετε ένα νεύμα διακριτικό με το χέρι στην καμπίνα 7. The second point is that this modification occurred only one month before the call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 Min revisor i Polen skrev til skat den 23. 4. 2009, og alt det blev sendt sammen med en klage på dansk fra min mands revisor, hvor vi har oversat noget af min revisors klage til dansk. Σας ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Έχουμε λάβει κάποιες απαντήσεις όσον αφορά την αφορά αυτή και το 2009 στείλαμε κάποια επιπλέον έγγραφα έγγραφα τα οποία πήγανε προς τις αρμόδιες φορολογικές αρχές. δεν λάβαμε απάντηση σε κανένα από τα αιτήματά μας αυτά. Λοιπόν, υπάρχει ένα συγκεκριμένο σχέδιο δράσης προκειμένου να προβλεφθεί ένα καθεστώς εξαίρεσης για το όχημά μου. Πρέπει να έρθει κανείς σε επαφή με την αρμόδια εθνική αρχή για να γίνει απαραίτητη ταξινόμηση του οχήματος αυτού. Και τα δύο μου αυτοκίνητα στα οποία αναφέρομαι αγοράστηκαν το 2009, ήρθανε οι απαραίτητοι ήρθαν οι αρμόδιοι από τις εθνικές αρχές για να μου πούνε ακριβώς ποια ήταν η διαδικασία που έπρεπε να ακολουθήσω, δεν έγινε σεβαστή η χρονική προθεσμία των 14 ημερών και οι εθνικές αρχές προχώρησαν στην κατάσχεση των οχημάτων. Εγώ από τη δικιά μου πλευρά δεν ήξερα τι έπρεπε να κάνω. Μου δώσανε απλώς την τελευταία στιγμή κάποιες πληροφορίες όσον αφορά το ζήτημα αυτό της ταξινόμησης. Χρειάστηκε στη συνέχεια να περιμένουμε έξι ολόκληρους μήνες και στη συνέχεια οι φορολογικές αρχές δεν απάντησαν. Είχαν μεσολαβήσει βέβαια και κάποιες, μια περίοδος διακοπών. έπρεπε να καταβάλω ένα τέλος ταξινόμησης για το πολωνικό μου αυτοκίνητο όντα στη Δανία. Αυτό το που μπορώ να σας πω είναι ότι ήρθα σε επαφή με όλους τους αρμόδιους όσον αφορά την υπόθεση αυτή και δεν είμαι η μόνη που βρίσκομαι στην περίπτωση αυτή. Υπάρχουν και άλλοι πολίτες πολωνικής ηθαγένειας που βρέθηκαν στην κατάσταση αυτή της κατάσχεσης του αυτοκινήτου τους, ενώ είχαν κάνει κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου να τακτοποιήσουν το θέμα της ταξινόμησης του αυτοκινήτου τους, το αυτοκίνητό τους ζώντας σε κάποια άλλη χώρα. Και εγώ που σας είπα προχώρησα σε όλες τις ε, ε, απαραίτητες ενέργειες όντας τη Δανία. Και μάλιστα δεν ήταν ιδιωτικής χρήσης το αυτοκίνητο αυτό, αλλά ήταν ένα αυτοκίνητο το οποίο μου είχε παραχωρήσει η επιχείρησή μου. Δεν μπορώ να καταλάβω λοιπόν για ποιο λόγο οι αρχές της Δανίας υιοθέτησαν τη στάση αυτή τη στιγμή που το αυτοκίνητο ήταν ένα αυτοκίνητο πολωνικής εταιρείας, το οποίο είχε ταξινομηθεί στην Πολωνία. Για ποιο λόγο πρέπει να γίνει μια αντίστοιχη ταξινόμηση και στη Δανία φαντάζομαι ότι η Δανία, όντα χώρα τη Ευρωπαϊκή Ένωση, υποχρεούται να προωθήσει την ελεύθερη κυκλοφορία και μετακίνηση των πολιτών. Για ποιο λόγο λοιπόν επιβάλλεται αυτό ο περιορισμό. Κάθε φορά που πηγαίνουμε στη Δανία θα πρέπει να προχωρούμε σε εκ νέου ταξινόμηση των οχημάτων μας. Θα θέλαμε λοιπόν να γνωρίζουμε τι πρέπει να κάνουμε όντας Πολωνοί πολίτες που ζούμε στην Δανία. Και τι πρέπει να κάνουμε στη συνέχεια προκειμένου να αντιμετωπίσουμε την κατάσχεση του οχήματο. Υπάρχουν και άλλοι Πολωνοί πολίτε οι οποίοι είχαν τέτοια προβλήματα όσον αφορά κατάσχεση από τις δανεικές αρχές ε, εταιρικού οχήματο. Πιστεύω λοιπόν ότι θα πρέπει να γίνει μια απαραίτητη εκστρατεία προτιθεί το πρόβλημα αυτό και οφείλω να σας πω ότι δεν μπορώ να καταλάβω για ποιο λόγο οι αρχές της Δανίας προχώρησαν στην κατάσχεση του εταιρικού οχήματός μου, όχι μόνο του πρώτου αλλά και του δεύτερου εταιρικού οχήματος. Ε, συγγνώμη, λέω για την ταχύτητα με την οποία μιλάω. Αν δεν κάνω λάθος, υπάρχουν συμφωνίες μεταξύ των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης Τέτοια συμφωνία υφίσταται στη Δανία εδώ και 25 χρόνια ιδανικές αρχές, ιδανική, ιδανικές αρχές αρμόδιες για τη φορολογία δεν δώσανε καμία βάσιμη δικαιολόγηση. Δεν γνωρίζω αν υπάρχουν και άλλες χώρες οι οποίες να αντιμετωπίζουν το ζήτημα της ταξινόμησης με αυτόν τον τρόπο. Με τις μεθόδους δηλαδή που ακολουθεί η Δανία. Καταλαβαίνετε ότι οι πολίτες επιβαρύνονται από πολλούς φόρους, από πολλά τέλη και το πρόβλημα είναι ότι μολονότι καταβάλουν τα τέλη αυτά, συνεχίζουν και αντιμετωπίζουν τα προβλήματα. Για ποιο λόγο λοιπόν θα πρέπει πάντα να πληρώνει ο Ευρωπαίος πολίτης, για ποιο λόγο να ζημιώνεται αυτός μόνο. Πρόκειται για οχήματα τα οποία εξαγοράστηκαν με νόμιμο τρόπο, προφανώς δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα προς αυτό. Θεωρώ όμως ότι δεν έγινε η απαραίτητη έρευνα και ότι δεν γίνανε σεβαστές όλες οι απαραίτητες διαδικασίες από τις δανεικές φορολογικές αρχές. Σε κάθε περίπτωση οι εργαζόμενοι στην ΣΚΕΤ έχουν ασχοληθεί εδώ και πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα με το ζήτημα αυτό. Δώσαμε προς το Υπουργείο Δικαιοσύνης όλα τα απαραίτητα έγγραφα τα οποία μας ζητήθηκαν, ζητήθηκαν. Γίνανε όλες οι προβλεπόμενες προσφυγές και αποφασίσαμε εν απουσία λύσης να απευθυνθούμε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μέσω της αναφοράς αυτής έχει ενημερωθεί τόσο η Πολωνία όσο και η Δανία, οι αρμόδιες αρχές δηλαδή στις χώρες αυτές. Συχνά αυτό το οποίο βλέπουμε είναι ότι ε, λαμβάνονται αποφάσεις χωρίς ε, να ακολουθούνται τα όσα προβλέπονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Πολύ συχνά υπερισχύει τελικά η εθνική νομοθεσία χωρίς να γίνεται σεβαστή η κοινοτική νομοθεσία. Φροντίσαμε πάντως εμείς να ενημερώσουμε και τα δικαστήρια της Δανίας, αποστέλλοντας όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Θα ήθελα να συνεχίσω κυρία Πρόεδρε, έχω να σας παραθέσω κάποιες ακόμα πληροφορίες Βλέπετε από το Σύνταγμα ότι τα πράγματα θα πρέπει να διεξάγονται με ένα ξεκάθαρο τρόπο. Βλέπουμε αυτή τη στιγμή ότι υπάρχει μια πολύ μεγάλη σύγχυση. Θα πρέπει εδώ πέρα να ξεκαθαριστεί ότι ε, η Δανία δεν εφαρμόζει την προβλεπόμενη κοινοτική νομοθεσία για το ζήτημα αυτό. Δίνω το λόγο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε.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 είναι τεχνικό πρόβλημα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ασχολήθηκε με το ζήτημα αυτό, άσκησε πίεση με αποτέλεσμα η Δανία να τροποποιήσει τους κανόνες της. Έκτοτε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρακολουθεί τους του σύνεγγε στην κατάσταση στην Δανία όσον αφορά την ταξινόμηση των οχημάτων και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θεωρεί πλέον ότι οι κανόνες που ακολουθεί η Δανία είναι οι κατάλληλοι, είναι οι σωστοί κανόνες. Επίσης, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενημερώθηκε ότι ο αναφέρον έλαβε το δικαίωμα να μπορεί να χρησιμοποιεί το εταιρικό του όχημα, το πολωνικό εταιρικό όχημα στην Δανία χωρίς να υποχρεούται να καταβάλει εκ νέου τέλος ταξινόμησης. Όσον αφορά την κατάσχεση οχημάτων που είναι ταξινομημένα σε άλλο κράτος μέλος, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ζήτησε από τη Δανία να αλλάξει την πρακτική την οποία ακολουθεί γιατί ε, ένα όχημα τέτοιου μεγέθους ταξινομημένο σε άλλο κράτος μέλος προφανώς οφείλει να μπορεί να κυκλοφορεί ελεύθερο στην ε, Δανία χωρίς πρόβλημα. Οι δανεικές αρχές όντως αναγνώρισαν ότι θα πρέπει να λάβουν δράση στον τομέα αυτό. Τροποποίησαν ήδη από τον Ιανουάριο κάποιους από τους κανόνες τους και υποσχέθηκαν να οριστικοποιήσουν την εσωτερική αυτή μεταρρύθμιση μέχρι το τέλος του μήνα. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας, κυρία Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Ούκεν. Να μιλήσω δανέζικα αυτή τη φορά. Πάρα πολύ ωραία. Ε, ήθελα απλά να πω ότι η απάντηση της Κομισιόν δεν είναι πλήρης, διότι Εάν η Δανία δεν σέβεται κάποιες αρχές, δεν είναι κάτι το οποίο μπορούμε να λύσουμε εμείς εδώ. Δεν είναι και αρμοδιότητά μας. Είναι θέμα, των, είναι θέμα νομικών διαδικασιών. Ε, και επομένως θα πρέπει να προχωρήσουμε κατά αυτήν την έννοια. Ο Σένθος Γιάρ. Μία ερώτηση θέλω να κάνω. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είπε ότι προφανώς η Δανία τροποποίησε Μάλλον όχι, αντιμετώπισε ε, ορθά τελικά το ζήτημα αυτό. Όμως φαίνεται ότι το πρόβλημα πλέον έχει διαλευκανθεί. Και αν αυτό ισχύει μπορούμε να κλείσουμε αυτήν την ε, αναφορά. Ε, και εν πάση περιπτώσει ε, οι φορολογικές, το φορολογικό δίκαιο αφορά τις χώρες μέλη. Δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι άλλο εμείς. και από τη στιγμή που βοηθήσαμε την αναφέρουσα, νομίζω ότι μπορούμε να κλείσουμε την αναφορά. Ένα λεπτό μόνο για να απαντήσει ο αναφέρον. Η τεκμηρίωσή μας καταδεικνύει ότι το νομικό σύστημα δεν άλλαξε και δεν εφαρμόζεται ακόμα το κοινοτικό δίκαιο. Απλώς ε, σε αυτή την περίπτωση βρέθηκε κάποια λύση. Πάντως δεν γίνεται σεβαστό το πνεύμα της ευρωπαϊκής νομοθεσίας. Είναι τρομερό αυτό που συμβαίνει στην ε, Δανία. Κατασχέσεις αυτοκινήτων, μεγάλα προβλήματα και για ανθρώπους πολιτικής καταγωγής και ε, για ανθρώπους πολίτες άλλων χωρών. Αυτό είναι παράλογο αυτό που συμβαίνει. Και δεν έχει καμία σχέση με την ε, σύζυγό μου για το που βρίσκεται ή που δεν βρίσκεται. Πουθενά δεν, ε, και καμία στιγμή η σύζυγός μου δεν έλαβε κάποια εξήγηση ή κάποια επιστολή. Όλες τα απαραίτητα στοιχεία τα έχουμε στείλει, αλλά κανείς δεν μας έχει δώσει οποιαδήποτε εξήγηση μέχρι τώρα. Δεν είναι δυνατόν ε, να μην ε, υπάρξει διευθέτηση του θέματος. Πρόεδρος, σας ευχαριστώ. Και πάντως η διαδικασία ακόμα εκρεμεί Άρα δεν μπορούμε εμείς να πάρουμε αποφάσεις γιατί βεβαίως εμείς είμαστε πάντα υποτελείς των εθνικών νομικών αρχών. Κάποιοι συνάδελφοι ζήτησαν να κλείσει η αναφορά. Όχι, κύριε, ο, ο, κύριος Γιάρ διορθώνει. Διάβασα την τελευταία πρόταση της απάντησης της Κομισιόν και λέει ότι η Κομισιόν θα παρακολουθήσει με προσοχή την εφαρμογή της κατευθυντήριας γραμμής μέσω των ε, αρμοδίων αρχών της Δανίας. Αυτή είναι μια πρόσφατη κατευθυντήρια γραμμή η οποία ικανοποιεί ιδιαίτερα την Κομισιόν. Αφήνουμε λοιπόν ανοιχτή την υπόθεση. Θα ήθελα να έχω μια απάντηση για να ξέρω εάν η εφαρμογή γίνεται ακριβώς με τον τρόπο από τον οποίο ε, θέλει η Κομισιόν. Ε, αυτή τη στιγμή ε, είναι δυνατόν οι αρμόδιες αρχές να παρέμβουν. Εγώ πιστεύω ότι η Δανία έχει αλλάξει κάτι, ε, ορισμένοι το αμφισβητούν, η εφαρμογή είναι αυτή που μας ενδιαφέρει, η κατευθυντήρια γραμμή είναι φρέσκια, πρόσφατη. Ας δούμε λοιπόν ε, τι θα μας πει η Κομισιόν, τις τελευταίες εξελίξεις και πώς θα μας ενημερώσει αν συνάδει η εφαρμογή με, με αυτά που επισημεί η Κομισιόν. Επομένως, θα αφήσουμε ανοιχτή την αναφορά μέχρι ότου μας κοινοποιήσει τη θέση, την στάση των Δανέζικων Αρχών ή Κομισιόν. Ωραία, θα περιμένουμε λοιπόν την απάντηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Επομένως μπορούμε να ολοκληρώσουμε τη συζήτηση από του σημείου αυτού και να περάσουμε στο επόμενο σημείο της ημερησίας διατάξεως, δηλαδή σημείο 17. Εκεί έχουν εγγραφεί τρεις αναφορές του Δαρίου Πατσάλα, του Άντωνη Μπιελάβα και του Γιάζεκ Ναγκουζεύσκη. Για τις τρεις αναφορές μονάχα ένας από τους ε, ε, υπογράφοντες ε, είναι παρόν, μονάχα δηλαδή ο Ρίζαρντ Άντωνη Μπιελάβα. Του δίνω αμέσω το λόγο. E, Ευχαριστώ. Έχω ζήσει στη Δανία τα τελευταία τρία χρόνια. Πριν από 18 μήνες κατασχέθηκε το αυτοκίνητό μου. Και εγώ συμμορφώθηκα με τις ε, απαιτήσεις των αρχών και ένα μήνα μετά την κατάσχεση και αφού είχα πληρώσει το πρόστιμο, πίστευα ότι θα έχω πάλι το αυτοκίνητο στη διάθεσή μου. Δύο εβδομάδες όμως αργότερα μου, μου στείλανε άλλη μια ιδιοποίηση για 25.000 κορώνες και το κόστος μεταφοράς του αυτοκινήτου 80 και 40 χιλιάδες κορώνος. <laughs> Δηλαδή, η αξία της μεταφοράς, τη δαπάνη της μεταφοράς του αυτοκινήτου ήταν περίπου δύο φορές η αξία του αυτοκινήτου. Η, η, φορολογική, ο ελεγκτής ε, μου είπε στην εφορία ότι αν δεν πληρώσω το ποσό αυτό θα έχω προβλήματα. Πράγματι, ρώτησα αν μπορώ να πληρώσω το πρόστιμο σε δόσεις και μου είπε ναι, 5.000 κορώνες ε, το μήνα λοιπόν συμφώνησα να πληρώσω και μου είπε ότι το αυτοκίνητο δεν θα απελευθερωθεί, αποδεσμευτεί, εάν δεν πληρωθεί όλο το πρόστιμο και εν συνεχεία μου είπε ότι πρέπει να πληρώνω και 3.000 κορώνες το μήνα για πάρκινγκ το πράγμα το οποίο βεβαίω δεν μπορούσα να κάνω γιατί ήμουν άνεργο. Εμείς ε, θέλαμε να φύγουμε από, την τη Δανία και να γυρίσουμε στην Πολωνία. Απλώ περιμένουμε να τελειώσει το σχολικό έτος για το παιδί μου και να φύγουμε από τη χώρα. Ε, άσχετο αυτό, αλλά εν πάση περιπτώσει είμαι τελείω αβοηθητο σε αυτή την ιστορία και υποστηρίζω την αναφορά 171 του 2010 διότι με μεταχειρίστηκαν ακριβώς με τον ίδιο τρόπο οι Δανέζικες αρχές. Ταξίδευα με την οικογένειά μου διότι ήμουν πολύ καιρό στο εξωτερικό, ταξίδευα από εδώ και από εκεί. Έφερα την οικογένειά μου στη Δανία για να μην χωρίσουμε ε, όπως είχαμε κάνει στο παρελθόν. Και ζητώ λοιπόν τη βοήθειά σας. Πλήρωσα τα, τις δαπάνες ε, καταχώρησης του αυτοκινήτου και όλα τα φιλόμενα και πρέπει να μου επιστρέψουν το αυτοκίνητο. Έχουμε αυτή τη στιγμή το σήμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης κολλημένο στο αυτοκίνητο. Ε, εδώ βρισκόμαστε μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι Δανείοι κάνουν ό,τι θέλουν και δεν εναρμονίζονται με τους υπόλοιπους. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ, Σουζάν Τάμς από την ε, Κομισιόν. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Θα ήθελα κι εγώ να μιλήσω για αυτή την, ε, ε, το, το, το, την υπόθεση που έχει τρεις πτυχές. Άσε, άσε. Και το αυτοκίνητο καταρχάς είχε καταχωρηθεί σε ένα άλλο κράτος μέλος και είχε ήδη πληρώσει ο αναφέρον το τέλος κυκλοφορίας εκεί, στη χώρα που είχε καταχωρηθεί το αυτοκίνητο. Μιλάω και για την 1444 αναφορά ταυτόχρονα. Εν συνεχεία, ε, ρώτησε εάν μπορεί να, ε, να καταχωρήσει το αυτοκίνητο και στη Δανία όσο καιρό δούλευε στη Δανία μαζί με την οικογένεια που ζούσαν μαζί δηλαδή και οι Δανικές αρχές είπαν ότι ο, εφόσον ο Πολωνός ε, ιδιοκτήτης του αυτοκινήτου έμενε στην Δανία θα έπρεπε να πληρώσει όλους τους φόρους και τους δασμούς και τα τέλη της Δανίας. Ε, υπάρχει λοιπόν μία νομολογία στη Δανία, αναπερίπτωση δεν υπάρχει σαφές ε, ή συγκεκριμένο νομοσχέδιο. Ε, Η νομολογία λοιπόν λέει ότι εάν μεταφερθείς από ένα κράτος μέλος σε ένα άλλο με την οικογένειά σου για να βοηθήσεις, για να δουλέψεις κατά ένα χρονικό διάστημα και δουλεύεις εκεί και εγκαθίσταται, τότε θεωρείται τόπος διαμονής. Και η Κομισιόν συμφωνεί με τις δανέζικες αρχές σε αυτή την περίπτωση, γι' αυτό εμείς δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Και συμφωνούμε με τις αρχές της Δανίας. Όμως, η διατύπωση των κανονισμών είναι τέτοια ώστε η, η, η είναι σωστή, η Κομισιόν τους ερμηνεύει ως σωστούς τους, τους κανόνες, τους κανονισμούς, αλλά όσον αφορά την κατάσχεση θα σχολιάσουμε αργότερα. Ευχαριστώ πολύ. Θέλουν οι συνάδελφοι να πούν κάτι. Ο κύριος Γιάρ, παρακαλώ. Μόνο ότι το θέμα αυτό είναι νομικό και δεν μπορούμε να βοηθήσουμε. Ε, είναι βεβαίως και το θέμα της ε, αναλογικότητας. Εάν οι φόροι δεν έχουν εναρμονιστεί, δυστυχώς ε, ισχύει η νομοθεσία του κράτους μέλους και δεν έχουμε καμία δυνατότητα να βοηθήσουμε ε, και παρά μόνο να εκφράσουμε την ε, δυσαρέσκειά μας για αυτή την κατάσταση, πιστεύω όμως ότι θα πρέπει να είναι ανάλογη η μεταχείριση του, της υπόθεσης, αναλογικότητα φόρων και δασμών. Νομίζω ότι εδώ είχαμε δύο περιπτώσεις και για εταιρικό αυτοκίνητο και για ε, προσωπικό ιδιωτικό αυτοκίνητο και η θέση μας είναι η ίδια. Ε, συμφωνώ με αυτά που λέει ο κύριος ε, Γιάρα, δηλαδή δεν υπάρχει λόγος ε, να αφήσουμε ανοιχτή την αναφορά, γιατί εμείς δεν έχουμε αρμοδιότητα περαιτέρω για το θέμα αυτό, άρα δεν θα έχουμε και καμία δυνατότητα παρέμβασης για να περιορίσουμε ας πούμε τις ζημίες που, κατακε... που καταγγέλλονται. Ένα λεπτό στον αναφέροντα για να απαντήσει. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε. Όπως είπα και προηγουμένως, εγώ ε, εγώ ακολούθησα την Δανέζικη νομοθεσία, πλήρωσα τους φόρους και δεν καταλαβαίνω γιατί δεν μου επιστράφει το αυτοκίνητο. Δεν το καταλαβαίνω γιατί εξακολουθεί η κατάσχεση. Ε, όταν πληρώνει κανείς αυτά που του ζητά το κράτος, θα πρέπει το κράτος να του επιστρέψει το αυτοκίνητο, γιατί εγώ εξαπατήθη, αισθάνομαι ότι έχω εξαπατηθεί. Ε, γιατί μου είπανε θα πληρώσεις το φόρο και μετά θα σου επιστρέψουν το αυτοκίνητο και το αυτοκίνητο δεν επιστράφει ποτέ. Πρόεδρος, ναι, προφανώς εδώ αυτό είναι μια απέτηση που αφορά αναγνώριση δικαιώματος για το οποίο όμως εμείς δεν, δεν έχουμε αρμοδιότητα. Ε, αυτό που μπορώ να φανταστώ είναι ε, να ε, ζητήσουμε ενδεχομένως κάποιες εξηγήσεις στις δανέζικες αρχές για την συμπεριφορά τους, δηλαδή να μας πούνε γιατί έχουν μια τέτοια αργή ανταπόκριση Ε, και επομένως ε, να τους ζητήσουμε όσο γίνεται πιο γρήγορα ε, να απαντήσουν, να ανταποκριθούν στα αιτήματα ανθρώπων όπως εσείς. Τώρα, εάν συμφωνούν και οι συνάδελφοι, μπορούμε να στείλουμε μια επιστολή στις δανέζικες αρχές, να τους παρουσιάσουμε εν συνθέσει όλες τις καταγγελίες οι οποίες, περι, οι οποίες περιέχονται στις αναφορές που μας απασχόλησαν και ε, να ζητήσουμε από τις δανέσικες αρχές ε, να κινητοποιηθούν πιο αποτελεσματικά έτσι ώστε ε, να υλοποιήσουν τις αποφάσεις οι οποίες ελήφθησαν. Αυτό θα κάνουμε και θα κλείσουμε τις αναφορές. Ευχαριστώ πολύ. Δεν μπορούμε να δώσουμε πλέον το λόγο για σε οποιονδήποτε γιατί ολοκληρώθηκαν αυτές οι αναφορές. Περνάμε στην αναφορά 18. Είναι η 590 του 2008. Ο αναφέρον δεν είναι παρόν αλλά η αναφορά έχει υποβληθεί από έναν ε, ε, Ιρλανδό υπήκο σχετικά με μεταφορά φαρμάκων ε, σε ταξιδιώτες που ταξιδεύουν στην Ευρώπη ο αναφέρον ε, διατείνεται ότι λόγω της ε, κατάστασης της υγείας του οφείλει να παίρνει μαζί του ε, φάρμακα και οι μεμονωμένες διατάξεις που αφορούν τη διακίνηση φαρμάκων, τη μεταφορά φαρμάκων στις ευρωπαϊκές χώρες του δημιουργούν προβλήματα. Ο κύριος Μωρίς Γκαλά από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ευχαριστώ. Αντικαθιστώ, δίνω το λόγο στη συνάδελφη που είναι ειδική. Ε, ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Πρόεδρε. Ε, ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε. Ε, μετά από την τελευταία μας επαφή το Μάιο του 2011, δυστυχώς δεν είχαμε καμία ενημέρωση σχετικά με, τα μέτρα τα οποία έλαβε η ε, Ιρλανδία για το θέμα αυτό. Ό,τι γνωρίζαμε ε, σας το έχουμε ε, δώσει. Μόνο την προηγούμενη εβδομάδα είχαμε ε, μια επιβεβαιωτική επιστολή από, το Ιρλανδικό Υπουργείο Υγείας. Δεν έχουμε τίποτα άλλο. Πρόεδρος, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θέλει κάποιος να πάρει το λόγο πάνω στο θέμα αυτό. Ε, ο, η γραμματεία μου λέει ότι και εμείς ελάβαμε μια επιστολή, ε, ανακοίνωση από την μόνιμη αντιπροσωπεία της ε, Ιρλανδίας επί του θέματος αυτού. Ε, και μπορούμε να μοιράσουμε στα μέλη της Επιτροπής την επιστολή αυτή. Δεν καταφέραμε να το κάνουμε ακόμα γιατί μόλις την λάβαμε. και επομένως ε, θα, να περιμένουμε ε, να ξανασυζητήσουμε την αναφορά όταν θα έχουμε λάβει γνώση του περιεχομένου των επιστολών αυτών. Συμφωνείτε πάρα πολύ, επομένως αφήνουμε ανοιχτή την επιστολή όταν ε, να μας ξανααπασχολήσει αργότερα θα έχουμε διαβάσει τις επιστολές. Σημείο 19 είναι η αναφορά 1665 του 2009 του Πίτερ Μπράουν, Βρετανικής Ιθαγένειας. Θα του δώσω το λόγο για 5 λεπτά, είναι παρόν ο αναφέρον. Thank you for inviting me. Um, Σας ευχαριστώ πολύ που με προσκαλέσατε. Η αναφορά μου είναι σαφέστατη Ε, θα, ε, στο σημείο μου που έχω στείλει αναφέρεται ότι θα έπρεπε να πληρώσω 5 εκατομμύρια ε, ευρώ, ή εγώ ή ο κατασκευαστής. Αυτό ήταν πάρα πολύ υψηλό ποσό και δυστυχώς καταγκάστηκα να κλείσω την επιχείρησή μου. Έπρεπε ο, η αναφορά και ο έλεγχος αυτός να έχει γίνει νωρίτερα και πιο εδελεχώς και πιο σωστός. Υπάρχουν ακόμα ε, καρκινογενείς ουσίες που κυκλοφορούν ελεύθερα στην αγορά για, ε, από, για τη, στη γεωργία, για λιπάσματα, για απολυμαντικά προϊόντα κλπ. Ε, Υπάρχει λοιπόν ένα εγγραφό, ένα φύλλο που αναφέρεται σε αυτές τις επικίνδυνες ουσίες, αλλά δεν είναι απαγορευμένες. Μπορεί να είναι επικίνδυνες, αλλά όχι απαγορευμένες. Είχα λοιπόν να απαντήσω σε πέντε ερατηματολόγια. Εγώ, ένα ήταν για τους χρήστες. Εγώ ήμουν χρήστης, δεν με ενημέρωσαν και εν συνεχεία το συμπέρασμα όλης αυτής της μελέτης ε, ρώτησα πόσο κόστισε και μου είπαν ότι το κόστος ήταν άσχετο με την ερώτηση που έθεσα. Εγώ όμως ήθελα να ξέρω πόσο κόστισε στους φιλουγούμενους μία μελέτη επιπτώσεων η οποία καταλήγει μόνο σε εικασίες. απευθύνθηκα στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Υπέθρου και μου είπαν ότι αυτά τα προϊόντα με υδροχλωρική στριχνίνη ε, είναι σταθερά προϊόντα και επίσης απευθύνθηκα σε γιατρούς που έχουν κάνει παρόμοιες μελέτες ε, στο Ηνωμένο Βασίλειο και μου είπαν ότι αυτή η ουσία είναι πιο αποτελεσματική για ε, αγροτικές ε, καλλιέργειες μεγάλης κλίμακας. Ο Βρετανικός Οργανισμός Ελέγχου των, ε, ζυζανιο, των Ζυζανιοκτώνων έκανε μία, τον παρασύρει Συντοκτόνων έκανε μία ε, έρευνα για την εξέταση αυτής της ουσίας ε, και αυτό βεβαίως επέφερε ένα κόστος. Ε, το όλο το κόστος όλων αυτών των μελετών το επιβαρύνθηκε ο φορολογούμενος. Όμως, δύο Γερμανοί εμπειρογνώμονες, οι οποίοι έκαναν αυτή την πρώτη μελέτη που σας είπα, κατέληξαν σε εικασίες και όχι σε συγκεκριμένα συμπεράσματα και ούτε ξέρω πώς κόστησε αυτή η μελέτη. Σας λέω όμως ότι στη γεωργία, σε αγροτικές καλλιέργειες ε, και για ε, τον έλεγχο των παρασίτων και ζυζανίων χρησιμοποιείται αυτή η ουσία για πάνω από 50 χρόνια. Λοιπόν, γιατί πρέπει εγώ να πληρώσω ε, τα λάθη των άλλων ε, όταν ε, μία υπηρεσία μου λέει ότι αυτή είναι επικίνδυνη ουσία, ενώ άλλες ε, επιτρέπουν τη χρήση εδώ και πολλά χρόνια. Σας είπα λοιπόν ότι η βελτίωση της νομοθεσίας θα μειώσει το κόστος. Σωστό, αλλά εγώ έχασα την επιχείρησή μου, όπως σας είπα, πριν από 5,5 χρόνια, καταστράφηκα δηλαδή και αναγκάζομαι να κάνω τρεις δουλειές τώρα για να τα βγάλω πέρα ενώ ταυτόχρονα χρησιμοποιούνται άλλες ουσίες που όχι μόνο είναι επικίνδυνες αλλά και παράνομες. Υπάρχουν παραθυράκια στην νομοθεσία. Ε, όλη αυτή η ιστορία ήρθε στην επιφάνεια πάρα πολύ αργά, με τεράστια ζημιά για μένα. Εγώ δεν έκανα τίποτα παράνομο, δεν ενήκησα κατά του νόμου ε, και δυστυχώς ε, τα μέλη έχουν ανεπαρκείς πληροφορίες ενώ, ενώ μου λένε ότι ε, εγώ έδωσα ανεπαρκείς πληροφορίες στα μέλη, δεν είναι σωστό αυτό, διότι όλες οι πληροφορίες ήταν στην αναφορά μου. Το συμπέρασμα είναι ότι αυτή η νομοθεσία με έχει διαλύσει, ε, υπάρχουν ε, γεγονότα πραγματικά στο περιβάλλον της γεωργίας ειδικά που δεν έχουν επιληθεί, υπάρχουν προβλήματα τα οποία υφίστανται ε, υπάρχουν αρχές οι οποίες δεν επιτελούν το έργο τους σωστά και αυτοί που είναι αρμόδιοι για την καταπολέμηση των παρασίτων, ζυζανίων κλπ. Ε, δεν έκαναν τη δουλειά τους και δεν εξέφρασαν την άποψή τους εγκαιρός. Γι' αυτό ακριβώς κάνω ε, μία αναφορά ε, στο Ευρωκοινοβούλιο ε, και μην ξεχνάτε ότι γίνονται δαπανηρές εκθέσεις για άλλες φαρμακευτικές ουσίες, το Viagra, το λοιπά χωρίς αντίρρηση. Θα ήθελα λοιπόν ή να με αποζημιώσετε ή να, με, προσαρμόσετε την νομοθεσία. Είπα, μου είπαν ότι θα γίνει μια διαρευνητική επίσκεψη. Πολύ ωραία ελάτε, ε, ελάτε, ε, επισκεφθείτε τις μονάδες, τις παραγωγικές μονάδες, δείτε την πραγματικότητα. Καταρχάς το κλίμα, μας, το κλίμα μας, όπως ξέρετε, είναι πάρα πολύ κρύο, αλλά εν πάση περιπτώσει ελάτε όποτε θέλετε. Αυτά. Ευχαριστούμε πολύ. John Benstel, Joan Benstel, από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Θα ήθελα να αναφέρθω κα... καταρχάς στις βασικές αρχές της οδηγίας. Uh, ε, αυτή λοιπόν η οδηγία για τα βιοκτώνα λέει ότι οι ουσίες αυτές είναι τοξικές για το περιβάλλον και για την υγεία, την ανθρώπινη υγεία και γι' αυτό τα βιοκτώνα αυτά μπορούν να, τεθούν, κυκλοφορήσουν στην αγορά μόνο εφόσον έχει γίνει η αξιολόγηση των ενδεχομένων κινδύνων. Ο στόχος λοιπόν αυτού του κανονισμού είναι να τονίσει ε, το, την προστασία της, του περιβάλλοντος και της ανθρώπινης υγείας. Η οδηγία προβλέπει μία αναθεώρηση και αξιολόγηση όλων των προϊόντων ε, των βιοκτώνων που χρησιμοποιούνται σήμερα. Μέσα στο πλαίσιο αυτής της αναθεώρησης η παραγωγική βιομηχανία βιοκτώνων έπρεπε να αναθεωρήσει όλα τα προϊόντα και τα, οι εταιρείε ε, οι οποίες χρησιμοποιούν ακόμα ενεργές ουσίες έπρεπε να κοινοποιήσουν τη χρήση τους και ποιες ουσίες. Ε, αυτό βεβαίως συνεπάγεται και την, ε, την συλλογή αλλά και αξιολόγηση όλων των στοιχείων που υποβάλλονται. Ε, η νομοθεσία λέει ότι εάν μια εταιρεία δεν δηλώσει ότι έχει την πρόθεση να υποστηρίξει μια ουσία, τότε η Κομισιόν παίρνει την απόφαση να, ε, μέσα σε μια εύλογη χρονική περίοδο, να απαγορεύσει την ε, χρήση της, του βιοκτώνου αυτού. Μία απαγόρευση λοιπόν δεν βασίζεται σε μία αυθαίρετη απόφαση, αλλά βασίζεται στο ότι δεν μπόρεσε να γίνει μία μελέτη αξιολόγησης του ενδεχόμενου κινδύνου. Αυτή η διαδικασία ισχύει για όλες τις ενεργές ουσίες ε, που χρησιμοποιούνται στην ευρωπαϊκή αγορά. Εάν δεν εφαρμόστηκαν αυτές οι, αυτοί οι κανόνες στην υδροχλωρική στριχνίνη, έγινε το εξής. Η ουσία αυτή υπήρξε στους γενικούς κανόνες, ταυτοποιήσει και ως βιοκτόνο δεν υπήρχε καμία εταιρεία, παραγωγός ή κυβέρνηση που δήλωσε ότι θα υποστηρίξει τη χρήση αυτής της ουσίας και που να υπέβαλε τα απαραίτητα στοιχεία. Ως αποτέλεσμα δεν έγινε καμία, δεν μπόρεσε να γίνει μελέτη αξιολόγησης κινδύνων και μαζί με άλλες ουσίες ή ε, στριχνίνη, η τροχλωρική στριχνίνη ε, έλαβε μία διάρκεια ζωής μέχρι το Σεπτέμβριο του 2006 και μετά από το Σεπτέμβριο του 2006 δεν θα μπορούσε πλέον να χρησιμοποιηθεί, θα ήταν απογορευμένη ουσία. Όπως είπε ο αναφέρον, το Ηνωμένο Βασίλειο ζήτησε μία παράταση της περίοδου ε, απαγόρευση. απαγόρευσης ε, η Κομισιόν ε, επέκταση δηλαδή αυτής της περίοδου μέχρι το Σεπτέμβριο του 2006 δεχτήκαμε την παράταση. Τώρα, οι πληροφορίες που λάβαμε ήταν εκ διαμέτρου αντίθετες. Ορισμένε πληροφορίες έλεγαν ότι η ουσία αυτή πρέπει να, επιτραπεί, να, πρέπει να επιτρέπεται να χρησιμοποιείται. Άλλοι λέγαν ε, που χρησιμοποίησαν άλλες παραδοσιακές μεθόδους όπως παγίδες κλπ. ότι η ουσία αυτή πρέπει να απογορευτεί. Και η απόφαση της Κομισιόν ήταν να διατηρηθεί η, περίοδο, η περίοδος αυτή του phase out, της βασμιάς απάλληψης δηλαδή, και στο διάστημα αυτό, καμία άλλη χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έδειξε ότι είχε σημαντικά προβλήματα ε, με την απαγόρευση της χρήσης, της τεχνίνης. Ε, τώρα, στα πλαίσια της αναθεώρησης ε, της οδηγίας των βιοκτώνων, που την ανέφερε ο, ο αναφέρον, η Κομισιόν πρότεινε μία αναθεώρηση για να μπορέσουμε να μελετήσουμε ορισμένα προβλήματα που εμφανίστηκαν με την εφαρμογή της οδηγίας. Το 2009 έγινε η νέα πρόταση της Κομισιόν βάσει μιας μελέτης επιπτώσεων του 2008 και η διαβούλευση των ενδιαφερομένων έγινε το 2006. Η διαβούλευση των ενδιαφερομένων ε, ξεκίνησε από την ιστοσελίδα της Γενικής Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και είναι ατυχές το ότι ο κύριος Μπράουν δεν μπόρεσε να συμμετάσχει και να συμβάλλει στην διαβούλευση αυτή Είχαμε όμως πολλές απαντήσεις και συμμετοχές άλλων ενδιαφερομένων για την ουσία αυτή. Η πρόταση της Κομισιόν του 2009 βασίζεται στην ε, ευελιξία που χρειάζεται για τη συλλογή και αξιολόγηση των στοιχείων και προσπαθεί να υποστηρίξει μικρομεσαίες επιχειρήσεις όμως ε, ο βασικός μας στόχος είναι ο ίδιος. Εμένουμε δηλαδή ότι πρέπει να εξασφαλίσουμε ένα υψηλό επίπεδο προστασίας του περιβάλλοντος και της ανθρώπινης υγείας με βάση των μελετών αξιολόγησης κινδύνου των βιοκτώνων. Και στην αρχή αυτή εμένουμε, δηλαδή ότι οι πληροφορίες της τοξικολογίας και της οικοτοξικολογίας, οι μελέτες αυτές δηλαδή τοξικολογικές, δεν θα πρέπει να είναι υπερβολικά μέσα στο πλαίσιο αυτό η Κομισιόν έχει ενεργήσει σωστά βάσει του, του νομοθετικού πλαισίου. Η Κομισιόν έλαβε όλα τα απαραίτητα μέτρα για να αξιολογήσει την εφαρμογή της οδηγίας και ανταποκρίθηκε σε ορισμένες ανησυχίες και προβλήματα που προέκυψαν. Ο κ. Μπράουν ρωτάει, μπορώ να μιλήσω. Ένα λεπτό λέει η πρόεδρος. Ένα λεπτό. Ο κ. Μπόλαντ. Σα Σας ευχαριστώ. Όσον αφορά το ζήτημα των βιοκτώνων και των ζυζανιοκτώνων, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει ορθή στάση εδώ. Δεδομένων των όσων λέει η οδηγία και δεδομένη της αρχής της πρόληψης. Ως προς αυτό λοιπόν θα ήθελα να πω στον αναφέροντα ότι συντοπίω τις δυσκολίες τις οποίες χρειάστηκε να αντιμετωπίσει από επαγγελματική πλευράς, αλλά θα πρέπει να γνωρίζουμε ότι είναι απόλυτα λογικό ότι με την πάρδα του χρόνου, μόλον ότι μπορεί στο παρελθόν να είχαν δοθεί κάποιες αδειοδοτήσεις για τη χρησιμοποίηση συγκεκριμένων ζανιοκτώνων, όπως είχαν δοθεί άλλωστε και αδειοδοτήσεις για να χρησιμοποιηθούν συγκεκριμένα φάρμακα κάποια εποχή Καταλαβαίνετε ότι ε, συνεχίζουμε και παρακολουθούμε συνεχώς τις επιπτώσεις που έχουν ορισμένα ζανιοκτώνα και φάρμακα στον άνθρωπο και στόχος μας είναι να δούμε αν υπάρχουν κάποιες επιθύμητες ενέργειες οι οποίες προκύπτουν και τις οποίες ενδεχομένως να μην είχαμε υπολογίσει στο παρελθόν, να μην τις είχαμε εντοπίσει. Εδώ και 50 λοιπόν χρόνια ανεχτήκαμε πάρα πολλά πράγματα όσον αφορά το περιβάλλον και όσον αφορά την ανθρώπινη υγεία, μέχρι που συνειδητοποιήσαμε ότι με τα τελευταία δεδομένα της επιστήμης υπήρχαν κάποιες επιζήμιες επιπτώσεις τόσο για τον άνθρωπο και το περιβάλλον. Συνεπώς, πιστεύω ότι θα πρέπει να υποστηρίξουμε περισσότερο την αρχή της πρόληψης και προς αυτήν πρόσκυμε τελικά περισσότερο. Και είναι σημαντικό βάσει αυτής να καθορίσουμε τις κυρώσεις ή τις επιζήμιες επιπτώσεις που βαρύνουν τελικά τους παραγωγούς ζυζανιοκτώνων και αν θα πρέπει να προβληθεί τελικά κάποιο σύστημα αποζημίωσης. Φαντάζομαι ότι η μελέτη αυτή πρέπει να εμβαθυνθεί λίγο περισσότερο, να μην επικεντρώνεται μόνο στη χρησιμοποίηση της υδροχλωρικής στριχνίνης κατά των αρουραίων. Είναι σημαντικό να γνωρίσουμε αν υπάρχουν κάποιες άλλες ουσίες που θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε, οι οποίες δεν θα ήταν επικίνδυνες. Ναι, ε, ο κύριος Γιάννη δεν θέλει, επομένως ε, ο αναφέρον για απάντηση. Ευχαριστώ πολύ. Συμφωνώ ότι βεβαίως θα πρέπει να κινούμεθα με προσοχή. Α, όμως στη Βρετανία επί πολλά χρόνια, επί δεκαετίες χρησιμοποιούσαμε ε, στριχνίνη. Για 60 χρόνια χρησιμοποιούσαμε την στριχνίνη. Είμαστε 40 χρόνια, είναι στη γνώση της Ευρωπαϊκής Ένωσης ότι χρησιμοποιούμε την ε, στριχνίνη. Ε, ξέρουμε ότι η στριχνίνη είναι θανατηφόρο ε, δηλητήριο. Δεν έγινε χθες θανατηφόρο δηλητήριο, ήταν από την αρχή και ήταν και εδώ και δεκαετίες γνωρίζει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ε, έχει συγκεκριμένα στοιχεία ε, σχετικά με την επίπτωση που μπορεί να ε, ε, έχει η δραστηριότητα αυτή με τη στριχνίνη είτε σε ανθρώπους είτε σε ζώα. Επίσης η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει σαφή ε, και ατράνταχτα επιστημονικά στοιχεία σχετικά με, την, με το ενδεχόμενο παρενεργειών στην ανθρώπινη υγεία αυτού του είδους της χρήσης της στριχνίνης. Ε, ε, ε, εδώ μας λένε ότι προκύπτει κίνδυνος για την ανθρώπινη υγεία από την μόλυνση των εδαφών. Εδώ όμως βλέπω ότι δεν υπάρχει κανένα τέτοιο, κανένα τέτοιο ενδεχόμενο. Ε, εδώ αναφέρεται απλώς ε, η περίπτωση κάποιων μορφών ασθενειών, αλλά αυτές οι ε, μορφές δεν συνδέονται με τη μόλις των εδαφών από τη χρήση της τριχνίνης, αλλά από επιζωτίες οι οποίες δεν έχουν καμία σχέση με αυτό. Εδώ και τρία χρόνια ασχολούμαι με το θέμα αυτό και με εκπλήσει ότι ε, ούτε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ούτε κανένας άλλος δεν έχει καταδείξει με τα βεβαιότητος την ύπαρξη κινδύνου. Δεν μιλάμε μονάχα βεβαίως για ανθρώπους, μιλάμε και για τα ζώα η στριχνίνη εδώ και 70 χρόνια χρησιμοποιείται στη, στο Ηνωμένο Βασίλειο ε, γιατί και, και ήταν ε, ε, σε, σε, μεγάλο ποσοστό ε, η, κυριότερη παγίδευση των ζώων και βεβαίως Ξέρετε ότι για τις παγίδες, η χρήση των παγίδων μπορεί να είναι πολύ αργός θάνατος ε, για τα ζώα ε, και μπορεί να πάρει και δύο και τρεις μέρες μέχρι να θανατωθούν. Ε, γι' αυτό λοιπόν νομίζω ότι θα πρέπει να δούμε λίγο από κοντά το θέμα αυτό. Η ε, νομοθεσία αυτή στην ουσία δημιουργεί μεγάλο πρόβλημα ε, και είναι επιζήμια για μεγάλα τμήματα του πληθυσμού. Γι' αυτό λοιπόν παρακαλώ να σκύψει πάνω στο θέμα αυτό η Επιτροπή σας. Ε, Πρόεδρος, νομίζω ότι η αναφορά αυτή έθιξε ένα ευαίσθητο ζήτημα. Θεωρώ ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν απήντησε ακριβώς στο συγκεκριμένο ζήτημα, αλλά ε, μας απεικόνισε την κατάσταση των πραγμάτων τούτη τη στιγμή, χωρίς όμως να δώσει την άποψη της Επιτροπής σχετικά ε, με την δυνατότητα ε, αναθεώρησης της οδηγίας ή μέσω άλλου τρόπου, την δυνατότητα λέγω, αντιμετώπισης ε, του συγκεκριμένου προβλήματος ε, το οποίο προκύπτει στα πλαίσια της ευρωπαϊκής νομοθεσίας. Νομίζω ότι σκόπιμο θα ήταν να ζητήσουμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή μια περαιτέρω προσπάθεια έτσι ώστε να έχουμε την ε, σωστή τεκμηρίωση η οποία θα καταδεικνύει ε, την ε, κατεύθυνση προς την οποία οδηγείται η Επιτροπή. Δηλαδή ε, θα αποφασίσει να κλείσει τελείως το θέμα ή θα αφήσει κάποια δυνατότητα να μείνει ανοιχτό έτσι ώστε ενδεχομένως να υπάρξει αναθεώρηση της υφιστάμενης και ισχύουσας οδηγίας. Θα ζητήσουμε λοιπόν αυτού του είδους την αποσαφήνιση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και δεν ξέρω εάν είναι δυνατόν η αποσαφήνιση αυτή να δοθεί σήμερα ή εάν θα μας στείλει κάποια γραπτή απάντηση. Στρέφομαι λοιπόν προς την εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Τι μπορεί να μας απαντήσει try respond quickly to your uh, request. Ευχαριστώ για να απαντήσω σύντομα στο έτοιμά σας. Καταρχάς, ε, σήμερα δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί πλέον. Όλες οι διαδικασίες έχουν εξαντληθεί από την υπάρχουσα οδηγία δεν λάβουμε από κανέναν κατασκευαστή, εταιρεία, χρήστη κλπ. ενδείξεις ότι θέλουν να υποστηρίξουν, να χρησιμοποιήσουν αυτή την ουσία. Ούτε υπάρχουν τα τοξικολογικά στοιχεία που να καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι αυτή η ουσία μπορεί να χρησιμοποιηθεί ακίνδυνα για βιοκτώνα. Όπως εξήγησε συνάδελφός μας, κάναμε μία εκτεταμένη αναθεώρηση της οδηγίας του 2006 και ξανά καταλήξαμε στο ε, συμπέρασμα ότι επειδή τη βάση όλων των στοιχείων και ενδείξεων που είχαμε για, εναλλακτικές, για χρήση εναλλακτικών ουσιών, προχωρήσαμε στην οριστική παύση χρήσης, απαγόρευση χρήσης αυτού, αυτής της ουσίας, εάν στο μέλλον προκύψουν καινούργια στοιχεία και συνταχθεί ένας νέος φάκελος υπέρ της χρήσης υδροχλωρικής τριχνίνης, τότε θα ξαναγίνει μία προσπάθεια, θα ξεκινήσει μία νέα προσπάθεια αλλαγή τη νομοθεσία επί τη βάση των νέων στοιχείων. Πάντοτε λοιπόν μπορεί να αλλάξει κάτι. Αλλά εμείς είμαστε υποχρεωμένοι πριν ε, συμπεριλάβουμε μία ουσία στις επιτρεπόμενες ουσίες, να έχουμε όλα τα τοξικολογικά στοιχεία, όλα τα απαραίτητα στοιχεία και δεδομένα στη διάθεσή μας για να μπορούν να ενσωματωθούν στην νομοθεσία. Ε, διαφορετικά δεν μπορούμε να κάνουμε μία μελέτη ε, αξιολόγησης κινδύνων. Δεν είχαμε τη δυνατότητα να κάνουμε αυτή τη μελέτη και έτσι αποσύρθηκε αυτή η ουσία. Αν όμως ξανά έρθει ένας πλήρης φάκελος με στοιχεία στα χέρια μας, θα ξαναγίνει μια νέα αξιολόγηση. Αυτά. Πρόεδρος, ε, δεν φαίνεται να θέλουν να παρέμβουν συνάδελφοι. Δεν υπάρχει περαιτέρω εμβάθυνση. Ο αναφέρον, συγγνώμη, αλλά δεν συμφωνώ. Όλα αυτά τα χρόνια, λέει ο κύριος Μπράουν, 60-70 χρόνια χρησιμοποιήθηκε στο Ενωμένο Βασίλειο, 40 χρόνια στην Ευρωπαϊκή Ένωση και δεν και αυτή τη στιγμή χρησιμοποιούνται άλλες ουσίες που είναι καρκινογενή αποδεδειγμένα με στοιχεία από τις Βρετανικές Αρχές, από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας κλπ. Και είναι στον κατάλογο επιτρεπόμενων ουσιών και χρησιμοποιείται παρόλο που είναι καρκινογενής αυτή η άλλη ουσία. Ενώ με τη στριχνίνη ε, πρέπει να επανεξεταστεί ο φάκελος, να ξανανοίξει ο φάκελος με όλα τα στοιχεία όλοι θα πρέπει να συμμετάσχουν στη διαβούλευση ελεύθερα και όχι μόνο να απαντούν σε κομμένα και ραμμένα, σε προετοιμασμένα ερωτηματολόγια. Ε, ε βασικά εφαρμόζουμε το, την αρχή της πρόληψης. Ε, κοιτάξτε, δεν είναι δυνατόν να δεχτούμε όταν μιλάμε για θέματα υγείας ε, τα ε, τέτοιου είδους συζητήσεις. Ε, δηλαδή δεν μπορεί να κάνουμε οικονομικές θεωρήσεις ε, όσον αφορά συγκεκριμένους στόχους, συγκεκριμένα στοιχεία τα οποία έχουν καταδειχθεί επιστημονικά. Δεν μπορεί να έχουμε οικονομικές θεωρήσεις για πράγματα τα οποία μπορούν να βλάψουν ε, την ε, υγεία. Τώρα το κατά πόσον η στρεχνίνη μπορεί να θεωρηθεί η βιοκτόνο ή εντομοκτόνο που μπορεί να διατηρηθεί, όπως είπατε κυρία Πρόεδρε, νομίζω ότι θα πρέπει να δούμε λίγο ε, τι γίνεται με την οδηγία για τα βιοκτόνα και να δούμε ποια είναι η κατεύθυνση που θέλει να πάρει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Πρόεδρος. Τώρα νομίζω ότι πια ε, δόθη εξαντλητική απάντηση, ε, έστω και αν δεν συμφωνεί ο αναφέρον με τα στοιχεία τα οποία έχουν υποβληθεί. Νομίζω ότι μπορούμε να κλείσουμε πλέον την αναφορά αυτή. Δεν έχουμε κάτι άλλο να κάνουμε, ε, αλλά βεβαίως να ε, υποβάλουμε αυτή την έκκληση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, να απαντήσει όσον αφορά την κατάσταση. Αλλά βεβαίως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή απήντησε και εδώ δεν φαίνεται να υπάρχει λόγος για περαιτέρω εμβάθυνση. Εν πάση περιπτώσει όμως εμείς δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι παραπάνω, επομένως νομίζω ότι θα συμφωνήσουν οι συνάδελφοι να κλείσουμε ε, την αναφορά δυστυχώς χωρίς να ικανοποιήσουμε ιδιαίτερα τον αναφέροντα. Περνάμε τώρα στο επόμενο σημείο της ημερησίας διάταξης. Είναι η αναφορά 500 του 2010 του Σαβέριο Ντεμπόνης. Ο αναφέρον είναι παρόν και επομένως θα του δώσω πέντε λεπτά έτσι ώστε να μας πει δύο λόγια σχετικά με αυτήν την αναφορά η οποία επανέρχεται. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε, ευχαριστώ και τα μέλη της Επιτροπής. Ε, εδώ βρισκόμαστε έτσι ώστε να ε, σχολιάσουμε ε, την αναφορά αυτή η οποία παρέμεινε ανοιχτή. Ποια είναι η θέση μας μπορούμε να πούμε ότι το ευρωπαϊκό ε, δίκαιο δεν εφαρμόζεται, δεν εφαρμόστηκε αφού ε, κάναμε μία πρώτη παρουσίαση στην ε, ε, Ιταλική Επιτροπή Αντιτράστα, Αντιμονοπολιακών Πολιτικών και μια και δεν είχαμε καμία εθνική αντιμετώπιση για τον Ιταλικό χώρο, συνεχίσαμε την προσπάθειά μας. Πέρα από τις πέρα από την πρώτη αναγνώριση ότι υπάρχει ένα πρόβλημα το οποίο κατεδείχθη στην ακρόαση. Οι Ιταλικές αρχές έστειλαν μια γνωμοδότηση, την οποία σας έχουμε στείλει και εμείς με τη σειρά μας, βάσει του άρθρου 22 του, 200, του νόμου 207, κοινοποιώντας στις αρμόδιες αρχές, τις υφιστάμενες ε, αρχές, ε, ε, προτείνοντας να υπάρξει μία προσαρμογή των κανόνων έτσι ώστε το σύστημα να προσαρμοστεί καλύτερα στον ευρωπαϊκό κανονισμό. Επί τούτου η Επιτροπή αναφέρθηκε ότι θα πρέπει να εφαρμοστούν ε, στην εκτροφή των κουνελιών οι κανόνες οι οποίοι αποφασίστηκαν σε ευρωπαϊκό επίπεδο. ξεπερνώντας ε, οποιαδήποτε διακριτική μεταχείριση. Επίσης να πω ότι έγινε υποχρεωτική και ε, η ε, η σφραγίδα και η σωστή ετικέτα πάνω στο ε, κρέας των κουνελιών. Αλλά αυτό σε δεύτερη ανάγνωση δεν έγινε γνωστή. Δεν έγινε αποδεκτή. παρόλα αυτά εξακολουθεί να υπάρχει μια πάρα πολύ κακή λειτουργία της αγοράς όσον αφορά ε, την ε, στρέβλωση του ανταγωνισμού ε, και από εκεί προκύπτει η ηθική και ηλική ζημία. Οι ιταλικέ αρχέ θα έπρεπε είτε να εφαρμόσουν τον κανονισμό είτε να ξεκινήσουν ε, μια ανακριτική ερευνητική διαδικασία. Τα κράτη-μέλη τη Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπορούν βάσει της αρχή της ε, χρηστή ε, και σωστή συνεργασία να διατηρήσουν μέτρα τα οποία ε, στην ουσία καθιστούν, ε, ε, καθιστούν ανενεργούς τους κανόνες του ορθού ανταγωνισμού. Επομένως, όλα τα όργανα του κράτους και του δημοσίου θα πρέπει να μην εφαρμόζουν εθνικές αρχές οι οποίες αντιτίθενται, έρχονται σε αντίθεση μάλλον με την, με την ευρωπαϊκή νομοθεσία. Είτε ε, μιλάμε για τον έλεγχο της αγοράς, είτε μιλάμε για τη διασφάλιση σωστού ε, ανταγωνισμού. Η Ιταλική κυβέρνηση θα έπρεπε να σταματήσει να εφαρμόζει αυτούς, τους, αυτά τα σημεία του Ιταλικού νόμου που αντιτίθενται ε, στην Ευρωπαϊκή Νομοθεσία και δεν θα έπρεπε να προσπαθήσει να επικεντρώσει την προσοχή της μονάχα ε, στις ετικέτες ε, και στη σήμανση του κρέατος. Βλέπουμε εδώ ότι διάφοροι επιχειρηματίες προσπαθούν να παραβιάσουν τους αντιμονοπολιακούς κανόνες ε, και ε, ε, έχουμε και την στάση των αρχών που είτε παραδέχονται την στάση αυτή είτε την ανέχονται και εν πάση περιπτώσει δημιουργούν στρέβλωση του ανταγωνισμού μεταξύ των επιχειρήσεων. Στην προκείμενη περίπτωση ή ε, ο κανονισμός ο οποίος αναφέρεται στη λειτουργία της αγοράς κρέατος κουνελιού που μας απασχολεί ε, μπορεί να προκαλέσει πολύ ε, αρνητικές επιπτώσεις και σίγουρα περιοριστικές, να έχει περιοριστικές επιπτώσεις οι αντιμονοπολιακές ε, πρακτικές, ε, συγγνώμη, οι μονοπωλιακές πρακτικές ε, θα έπρεπε οπωσδήποτε να αποτελούν αντικείμενο κυρώσεων. Γνωρίζουμε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προσπαθεί ε, να ασχοληθεί με, τις, ε, με τους περιορισμούς που έχουν μεγαλύτερη οικονομική επίπτωση και δεν πολύ ασχολείται με θέματα τα οποία μπορεί να έχουν λιγότερο αντίκτυπο. Αλλά μικρότερος αντίκτυπος δεν μπορεί να σημαίνει ότι αφήνουμε ανοιχτές τις πόρτες για παραβίαση των ε, ευρωπαϊκών ε, κανόνων και των ευρωπαϊκών ε, νόμων. Και σίγουρα δεν μπορεί να επιτρέψουμε την παραβίαση των κανόνων του ελεύθερου ανταγωνισμού. Ζητούμε λοιπόν να ενεργήσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή βάσει της αρχής της επικουρικότητας η διαδικασία αυτή τη στιγμή δεν εκκρεμεί ενώπιον των Ιταλικών αρχών. Ζητούμε πάντως από την Ευρωπαϊκή Ένωση, ε, να, από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, να ξανακινήσει την διαδικασία έτσι ώστε να σταματήσει η παραβίαση από πλευράς των Ιταλικών αρχών. Θα πρέπει να διασφαλιστεί επομένως η σωστή εφαρμογή των κανόνων του ανταγωνισμού. Σύμφωνα με τις σύμφωνα με τις αρχές της Ευρωπαϊκής ε, ε, Επιτροπής ε, μπορεί να ξανανοίξει ένα ζήτημα εάν δεν έχουν ξεπεραστεί, δεν έχει ξεπεραστεί το διάστημα των δύο μηνών από την, από, την αρχή της ερευνητικής διαδικασίας. και ε, σε περίπτωση μονάχα που μπορεί να υπάρξει η άρση της ε, παραβίασης ε, γιατί μονάχα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μπορεί να κινηθεί προς αυτή την έννοια. Η Ένωσή μας έχει ήδη δώσει τα απαραίτητα στοιχεία στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή καθώς επίσης και στην ανακοίνωση που έκανε προς τα μέλη της Επιτροπής αναφέρθηκε σε όλα τα στοιχεία. Όμως εδώ ε, φαίνεται σαφώς ότι οι πράξεις δεν ακολουθούν τα λόγια και ότι δεν εφαρμόζεται το κοινοτικό δίκαιο. Ε, δεν είναι δυνατόν να θεωρήσουμε ότι η τροποποίηση της τιμής είναι αποτέλεσμα λογικών διακυμάνσεων της αγοράς και στον καθορισμό, ο καθορισμός των οικονομικών αρχών ε, μπορεί να δημιουργήσει μεγάλο πρόβλημα στους εκτροφείς των κουνελιών. Ε, σε αυτό ε, προστίθεται η δυσκολία, προστίθεται η ζημία των καταναλωτών διότι οι μειώσεις ε, τιμών δεν ε, ε, προκύπτουν και επομένως δεν προκύπτει και κάποιο όφελος για τους πολίτες της Ευρώπης. Θεωρούμε λοιπόν ότι θα πρέπει η τιμή να είναι τέτοια, η οποία, να είναι τέτοια που να αποδεικνύει ότι γίνονται σεβαστοί οι κανόνες του ανταγωνισμού και δεν μπορεί να περιοριστεί η προστασία των καταναλωτών μονάχα στην ετικετούλα με, το, με την ε, αναφορά της τιμής που θα ε, υπάρχει πάνω στο ε, κρέας. Και στο άρθρο 1 παραγραφός 6 διαφαίνεται σαφώς ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρέπει να παρακολουθεί την εφαρμογή του ευρωπαϊκού ε, δικαίου. Ε, ζητούμε λοιπόν η Ευρωπαϊκή Αντιμονοπολιακή Αρχή ε, να δράσει βάσει του άρθρου 101 της Συνθήκης Λειτουργίας Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ζητούμε να μείνει η αναφορά ανοιχτή μέχρι ότου έχουμε την σωστή απάντηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Επιτροπής. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ. Δεν έχουμε όμως εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, εδώ από την Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού. Έχουμε όμως τον Δόκτωρα Φλόιντ, ο οποίος ενδεχομένως ε, θα μπορούσε να μας πει δύο λόγια. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ζητώ συγγνώμη εξ ονόματος του συναδέλφου μου, ο οποίος έχει ασθενήσει, δεν μπορεί να είναι μαζί μας σήμερα. Θα ήθελα να υπενθυμίσω στην Επιτροπή σας ότι τέτοιες αναφορές στην αυτή την έχουμε δει και στο παρελθόν. Δηλαδή κάθε φορά που έχουμε να κάνουμε με θέματα ανταγωνισμού. Υπάρχει μια κατανομή δραστηριότητας ανάμεσα στις εθνικές αρχές ανταγωνισμού και τις ευρωπαϊκές αρχές ανταγωνισμού. Και το έχουμε εξηγήσει αυτό πολλές φορές στο παρελθόν εξετάζοντας αναφορές, ότι υπάρχουν τρία κριτήρια τα οποία θα πρέπει να ισχύουν προκειμένου να μπορούμε να κρίνουμε αν τελικά η αρμόδια αρχή είναι η εθνική αρχή ανταγωνισμού. Το πρώτο κριτήριο είναι οι επιπτώσεις αυτές να έχουν εθνική διάσταση. Δεύτερον, ότι θα πρέπει η Εθνική Αρχή Ανταγωνισμού να έχει την απαραίτητη αρμοδιότητα προκειμένου να διορθώσει την κατάσταση και τρίτον, η Εθνική Αρμόδια, η Εθνική Αρμόδια Αρχή για τον Ανταγωνισμό θα πρέπει να έχει τα απαραίτητα στοιχεία προκειμένου να ασχοληθεί με την υπόθεση αυτή. Στην περίπτωση αυτή, καταλαβαίνω βέβαια τι μας είπε ο αναφέρον, αλλά τα κριτήρια αυτά καταδεικνύουν τελικά ότι είναι εσωτερική υπόθεση της Ιταλίας το όλο ζήτημα εξακριβώσαμε ότι όντω ε, η, Ιταλική ε, διοίκηση ασχολείται με το ζήτημα αυτό. Αυτό φαίνεται και από την αρχική μα συμβολή στην υπόθεση αυτή. Επομένω, ε, αυτά μπορούμε να πούμε όσον αφορά το ζήτημα του ανταγωνισμού. Ο αναφέρον αναφέρθηκε και σε δύο άλλα ζητήματα. Στην ετικετοθεσία. Η Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, νομίζω ότι λίγο νωρίτερα αυτό το μήνα, ασχολήθηκε με το ζήτημα αυτό και όντω ήταν πολύ δύσκολο να βρεθεί μια συμβαστική θέση μαζί με το Συμβούλιο για το τι θα πρέπει να συμπεριλαμβάνεται στην ετικέτα και τι όχι. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αποφάσισε να ακολουθήσει τον υφιστάμενο συμβασμό και έτσι έχουν τα πράγματα αυτή τη στιγμή. Μία άλλη σημαντική πτυχή είναι ότι είναι πολύ σημαντικό να παρακολουθούμε την εξέλιξη των τιμών. Υπάρχει ένα παρατηρητήριο για, το, για τις τιμές, όχι μόνο για το κρέας, αλλά και για τα γαλακτοκομικά προϊόντα. Καταλαβαίνετε ότι στις αγορές αυτές η διάρθρωση είναι τέτοια που είναι πολύ δύσκολο πολλές φορές να γίνουν οι απαραίτητες διαπραγματεύσεις για την κατάρτιση των τιμών. Έχουμε ήδη τα πρώτα αποτελέσματα από τη δημιουργία αυτού του παρατηρητηρίου και είναι αυτή ουσιαστικά, αν θέλετε, σημαντικότερη συμβολή από τη δική μα την πλευρά, προκειμένου να δημιουργηθεί ένα υψηλότερο επίπεδο διαφάνεια στην διατροφική αλυσίδα, ιδίω όσον αφορά το ζήτημα των τιμών. Αυτέ τι πληροφορίε μπορώ να δώσω προ τα μέλη τη Επιτροπή σα σε αυτή τη φάση. Ευχαριστούμε πολύ. Ο κύριος Γιάρ θέλει να πει δύο λόγια. Ε, επειδή όλους μας εκνευρίζει αυτή η κατάσταση, ιδίως όσον αφορά τα προϊόντα για τα αγροτικά προϊόντα, τις τιμές για τα αγροτικά προϊόντα, θα ήθελα να θέσουμε το θέμα αυτό υπόψη και στην Επιτροπή Γεωργίας. Αυτό το οποίο βλέπω εγώ να γίνεται είναι ότι υπάρχει μία δομή μονοπωλιακή, ένα καρτέλ δηλαδή, το οποίο κανονίζει τις τιμές αντίθετα προς το συμφέρον των καταναλωτών. Δεν καταλαβαίνω πώς γίνεται αυτό. Ο εκπρόσωπος της ε, Κομισιόν είπε ότι οι τιμές που προσφέρονται στους παραγωγούς διακυβεύουν την επιβίωσή τους οι εμπορικές, ε, οι εμπορευόμενοι των προϊόντων αυτών είπαν ότι έχουμε αυτές τις χαμηλές τιμές για να εξυπηρετήσουμε τον καταναλωτό. Ναι, εντάξει, αλλά τι γίνεται με τον παραγωγό. Τώρα η όλη δομή των τιμών και πώς, το πώς διαμορφώνονται οι τιμές οδηγούν εν τέλει στην εξαφάνιση των παραγωγών και των εκτροφέων. Ε, πιστεύω ότι η αναφορά αυτή πρέπει να μείνει ανοιχτή, να τεθεί υπόψη της Επιτροπής Γεωργίας για γνωμοδότηση. Πρόσφατα έχει ασχοληθεί η Επιτροπή Γεωργίας ε, με το γάλα, αλλά γιατί να μην ασχοληθεί και με τα κουνέλια. Για γνωμοδότηση, ναι. Ε, allora, c'è qual... c'è una... Πρόεδρος. Ένα λεπτό σας παρακαλώ γιατί πρέπει να κλείσουμε. Στις παρατηρήσεις ε, της Επιτροπής ε, αναφέρθηκαν τρία κριτήρια, κυρίως δε ε, πρέπει να πω ότι οι συμφωνίες εξακολουθούν να προκαλούν αρνητικές επιπτώσεις στον ανταγωνισμό στην Ιταλική επικράτεια. Και σε μία υπόθεση η οποία παρά τις αντιτιθέμενες ε, απόψεις ε, αρχιοθετήθηκε. Ανεφέρεται ακριβώς το συγκεκριμένο θέμα ότι ενδεχομένω υπάρχει δηλαδή πρόβλημα. Ε, Πρωτοβάθμιο το δικαστήριο αποφάσισε ότι οι αντιμονοπολιακοί κανόνες δεν εφαρμόζονται και ότι η κατάσταση στη Γεωργία διαφεύγει του ελέγχου των αρχών γιατί στην ενδιάμεση φάση μεταποίησης ε, αυτή η ενδιάμεση φάση μεταποίησης και προώθησης στην αγορά στην ουσία υποκλέπτουν από τους ε, εκτροφείς ένα μεγάλο μέρος ε, του ελέγχου της αγοράς καθώς επίσης και του ελέγχου των τιμών. Νομίζω ότι παρά να προσπαθούμε να απευθυνθούμε στο πρωτοδικείο ή στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο θα πρέπει να καταλάβουμε τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν οι αντιμονοπολιακοί κανόνες. Ευχαριστώ πολύ. Έχουμε την πρόταση του συναδέλφου Γιάρ, δηλαδή να ζητήσουμε γνωμοδότηση από την Επιτροπή Γεωργίας όσον αφορά το τμήμα της αρμοδιότητας και νομίζω ότι όλοι συμφωνούμε γι' αυτό. Εγώ θα ήθελα να προσθέσω και κάτι άλλο, να προσθέσω μια άλλη πρόταση δηλαδή για το σκέλος το οποίο αφορά ε, τον ανταγωνισμό. Έχουμε ένα πρώτο στοιχείο. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δηλώνει ότι δεν μπορεί να παρέμβει περαιτέρω γιατί αυτή τη στιγμή ασχολείται με το θέμα ε, η Εθνική Αρχή και σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στο υπόμνημα της Επιτροπής από τη στιγμή που μία αρχή ε, από αυτές που συνεργάζονται στο Ευρωπαϊκό Δίκτυο Ανταγωνισμού δεν μπορεί να παρέμβει. Όμως ε, ο αναφέρον μας λέει ότι η διαδικασία αυτή, η οποία ακόμα εκκρεμεί ενώπιον των δικαστηρίων, ε, σε ολοκληρώνεται. Άρα δεν θα υπάρχει πρόβλημα μη αρμοδιότητας. Επομένως θα ζητήσω και από από την Εθνική Αρχή Ανταγωνισμού ε, ε, να μου πιστοποιήσει ότι όντω ολοκληρώνεται η διαδικασία η οποία εκκρεμεί ενώπιον του τελικού δικαστηρίου ε, και μετά να ζητήσω με την Επιτροπή να ασκήσει τις αρμοδιότητές της. Μπορώ να υπογραμμίσω ότι δεν είναι δυνατόν να δεχτούμε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν έχει λάβει καμία, καμία καταγγελία μέχρι σήμερα από την ΑΛΑΚ γιατί αυτού του είδους αυτού του είδους ε, οι δηλώσεις ε, στην ουσία ε, καταδεικνύει ότι η Επιτροπή δεν δίνει δεκάρα τσακιστή για, τα, για τις καταγγελίες που κάνει η δικιά μας Επιτροπή Αναφορών. Και εγώ μπορώ να σας διαβεβαιώσω ότι εδώ και ένα χρόνο τουλάχιστον η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έλαβε μέσω της δικής μας Επιτροπής ε, την καταγγελία αυτή. Επίσης, θα προσθέσω ότι θα στείλω και υπόμνημα στον Ιταλό Υπουργό Γεωργίας γιατί υπάρχουν και στοιχεία τα οποία αφορούν την αρμοδιότητα των εθνικών, του, του Εθνικού Υπουργείου Γεωργίας, κυρίως όσον αφορά τον ανταγωνισμό. Firmatario, da quello che abbiamo letto, non sembrano coerenti fino in fondo. Ε, και επομένως εξακολουθούν να παραμένουν στοιχεία ανοιχτά ε, και μπορώ να πω ότι εάν συμφωνείτε όλοι μπορούμε να αφήσουμε ανοιχτή ε, την αναφορά και να προχωρήσουμε με αυτές τις τρεις επιστολές τις οποίες ανέφερα, τρεις επαφές που ανέφερα. Όσον αφορά τώρα το σημείο ε, για την ετικετοθεσία. Ε, όντως το παρατηρητήριο τιμών είναι σημαντικό, αλλά ακόμα περιμένουμε να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες όσον αφορά τις ετικέτες. Ε, ήταν λίγο με ανδρόδηση η διαδρομή των ετικετών. Το γνωρίζουμε πολύ καλά ποιες διαδικασίες έτσι δύσκολες ε, ακολουθήθηκαν και είναι ένα πρόβλημα το οποίο δεν αφορά μονάχα τους κονικλόπαραγωγούς, είναι ένα γενικότερο ζήτημα. Ε, και νομίζω ότι και από αυτού η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα κληθεί ε, ξανά να απαντήσει. μπορούμε να στείλουμε ενδεχομένως και επιστολή άμεσα στον Επίτροπο Υπεύθυνο για θέματα ανταγωνισμού. Συμφωνείτε. Άρα τέσσερις οι επιστολές. Ναι, τέσσερα τα αιτήματα. Συμφωνείτε. Σας φαίνεται υπερβολική αυτή η προσέγγιση. Αλλά βλέπω ότι νεύεται καταφατικά και επομένως ωραία τέσσερις ε, λοιπόν ε, τετραπλή κοινοποίηση έτσι ώστε να είμαστε σίγουροι ότι η καταγγελία της Άνλακ θα φτάσει άμεσα και στα αυτιά του Επιτρόπου που είναι υπεύθυνο για τα θέματα ανταγωνισμού. Ολοκληρώσαμε λοιπόν την συνεδρίασή μας. Ε, βεβαίως είναι και η τελευταία συνεδρίαση αυτής ε, της ε, σχολικής χρονιάς αν μου επιτρέπετε να ευχηθώ καλές διακοπές σε όλους, στους βουλευτές, στους συνεργάτες, στους διερμηνείς. Ευχαριστούμε πολύ.